Ladies Κυρίες ε, και κύριοι, καλημέρα σας. Ε, πρωί πρωί, αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα. Τι να κάνουμε. Έχουμε μεγάλη συνεδρίαση μπροστά μας ε, και είναι ευχαριστησή μου να σας καλωσορίσω σήμερα στην δεύτερη ημέρα της συνεδρίασής μας. Σας ευχαριστώ. το επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης είναι κοινή συνεδρίαση με την Επιτροπή Εξωτερικών και χαιρόμαστε που έχουμε εδώ πέρα τον αντιπρόεδρο της Επιτροπής μας ο οποίος ε, θα κάνει και τις εισαγωγικές του παρατηρήσεις ε, και αυτό είναι επίσης συνεργασία με την αντιπροσωπεία του Κοινοβουλίου για τις σχέσεις ε, με το Παναφρικανικό ναι. Κοινοβούλιο και θα ήθελα να καλωσορίσω την αντιπροσωπεία Αφρικανών βουλευτών που συμμετέχουν στην διάσκεψη υψηλού επίπεδου του Προέδρου Ταγιάννη για τις σχέσεις ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, και Αφρικανικής Ένωσης. Σε λίγες μέρες ε, θα πάμε και εμείς στο Αμπιτζάν για την κοινοβουλευτική διάσταση της ε, Συνόδου Κορυφής ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης και βεβαίως ε, σωστό είναι να κάνουμε και μια συνεδρία σήμερα να δούμε όλα αυτά τα πράγματα και τις εκδηλώσεις κυρίως που σχετίζονται με την ε, πολύ σημαντική σύνοδο. Το θέμα μας εδώ είναι πολύ συγκεκριμένο. Αφορά την αποστολή Σαχέλ Μαλή, την αποστολή αυτή της ε, ΚΕΠΑ που έχει αναπτυχθεί εκεί και τον ρόλο αυτής της ε, αποστολής Νίγηρα ε, βεβαίως εννοούσα όχι Μαλή για να ενισχύσει τις ε, ικανότητες ε, της χώρας στην καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Πριν περάσω στις συστάσεις θα ήθελα να ζητήσω από τον αντιπρόεδρο της ε, ΑΦΕΤ να κάνει και αυτό στις ε, παρατηρήσεις του. ευχαριστώ Άννα. Θα ήθελα από τη δική μας την Σκοπιά να τονίσω την σημασία του Σαχέλ για την σταθερότητα και την ασφάλεια όλης της υποσαχαρίας Αφρικής αλλά και παραπέρα μέχρι και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Νομίζω πως είναι μια πολύ επίκαιρη συζήτηση και ακούσαμε διάφορα πράγματα και για το Σαχέλ και για την ανάγκη να διασφαλίσουμε την ειρήνη στην περιοχή εκεί και σε ολόκληρη την Αφρική Ακούσαμε τα όσα συμβαίνουν, τα οποία επηρεάζουν και την Ευρώπη με τον έναν τρόπο ή τον άλλον. Γι' αυτό η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει στην περιοχή. Λοιπόν, να σας ξαναδώ στον λόγο κυρία Πρόεδρε για να παρουσιάσετε τους προσκεκλημένους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρώτα απ' όλα λοιπόν να σας παρουσιάσω τον κύριο Μπέρτ Φερσμέσεν υποδιοικητής ε, μη στρατιωτικών επιχειρήσεων ε, και προσωπάρχης ε, της ΕΙΕΔ και βρίσκεται σήμερα μαζί μας κατόπιν Έχουμε έναν προσκεκλημένο από την χώρα, βεβαίω την ίδια, τον κύριο Μοχάμεντ Ανακό, τον περιφερειάρχη του Αγκαντέζ. Πολύ σημαντικό το θέμα αυτό και περιπεπλεγμένο από πλευράς ασφαλείας. Η αποστολή μας κατάφερε να δημιουργήσει μια προκεχωρημένη βάση στο Αγκαντέζ και βεβαίω γι' αυτό χαιρόμαστε που έχουμε εδώ πέρα και τον Περιφερειάρχη και τέλος έχουμε τον κύριο Άντριου Λέμποβιτς, εταίρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ε, Διεθνών Σχέσεων. Χωρίς ε, περαιτέρω καθυστέρηση λοιπόν ε, θα ήθελα να δώσω τον λόγο στα μέλη του πάνελ μας. Ξεκινάμε με τον κύριο Φερσμέσεν. La euh, Ευχαριστώ πολύ. Εκπροσωπώ τον κύριο Κέντιν που είναι στο Ιράκ αυτή τη στιγμή και τον ε, εκπροσωπώ εγώ. Το Ιράκ είναι ένα θέμα που θα σας απασχολήσει στη συνέχεια. Το Μάρτιο είχε έρθει στην Επιτροπή σας για να μιλήσει για την κατάσταση στο Σαχέλ και το σχέδιο περιφερειακής ολοκλήρωσης. Χαίρομαι που συμμετέχω στη συζήτηση αυτή. Πιστεύω ότι θα υπάρξει προσεχώς κοινή αποστολή ΑΦΕΤ που θα μεταβεί στον Ήγηρα. Όπως είπατε, Πρόεδρε, είναι πάρα πολύ ειδικό το θέμα για να ε, αναλύσουμε τι κάνει αυτή η αποστολή. Είναι μια πολιτική αποστολή, ΟΚΑΠ, την οποία ζήτησε η κυβέρνηση του Νιγηρά και αναπτύχθηκε το ε, θέρος του 2012 και συνιστά ένα στοιχείο στρατηγικής Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Σαχέλ, ε, για την ασφάλεια και την ανάπτυξη της περιοχής. Είναι μη εκτελεστική εντολή της και περιφερειακή η αποστολή της. Βασικό σκέλος δραστηριοτήτων είναι η Συμβουλή παροχή συμβουλών και ενημέρωσης για να ενισχυθούν οι ικανότητε ιστορικής ασφάλειας στον Ήγηρα. Να σας δώσω κάποια στοιχεία βασικά. Η κυρία Κίρση Χέριξον είναι επικεφαλής από το Σεπτέμβριο. Όπως σας είπα, η αποστολή ε, μετέβηκε το 2012 και η εντολή της ε, λεκπνέει τον Ιούλιο του 2018 με μια στρατηγική αναθεώρηση τον Ιανουάριο του 2018 αυτή τη στιγμή απαρτίζεται από 136 μέλη. 95 διεθνείς, ε, εξωτερικοί και 41 ντόπιοι. Στην ΙΕΜΕΗ είναι, ε, η έδρα και έχει και παράρτημα στο Καντές που ε, άνοιξε τον Απρίλιο του 2016. Ποιες είναι οι βασικές της υποχρεώσεις. Να υποστηρίξει τη διαλειτουργικότητα των δυνάμεων ασφαλείας ε, του Νιγήρα που είναι η αστυνομία, ε, η χωροφυλακή και η εθνοφυλακή. Να ενισχύσει τις τεχνικές ικανότητες και δυνατότητες των σωμάτων ασφαλείας, ε, κατάρτιση ανθρωπίνου προσωπικού, διαχείριση υλικού, υποστήριξη και πολύ σημαντικό ε, του διεθνούς και ε, περιφερειακού συντονισμού. Αυτά όλα ξεκίνησαν το 2012. Το 2015 άλλαξε η, η εντολή ε, για να βοηθήσει τις δυνάμεις ασφαλείας να καταπολεμήσει την παράτυπη μετανάστευση και τις εγκληματικές ενέργειες που συνδέονται με αυτή. Υπό τη σημερινή εντολή δίνεται με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια του Αγκαντές στο βορρά γιατί ε, είναι εκείνη που υφίσταται τις μεγαλύτερες απειλές για την ασφάλεια από την παράτυπη μετανάστευση και τα σχετικά λαθρεμπόρια. 20 φορές έχουν μεταβεί εκεί ε, για να εκπαιδεύσουν τα σώματα ασφαλείας, για να αξιολογήσουν τις ανάγκες και ενδεχομένως να δώσουν και εξοπλισμό. Για παράδειγμα, η αποστολή πρόσφατα πήγε στον Τύρκου, στο βόρειο ανατολικό Νίγηρα και στο Μάνταμα, κοντά ε, στα σύνορα με τη Λιβύη και στο Ζίνγκερ που είναι στη νότιο-δυτική περιφέρεια της χώρας πάντα σε συντονισμό με τις αρχές του, Νίκη, του Νίγηρα και δεν σας κρύβω ότι κάθε φορά αυτό είναι ε, μεγάλη δυσκολία από πλευράς επιμελητίας. Η τελευταία επίσκεψη έγινε σε συνεργασία με τη Frontex και την ε, Ευρωπαϊκή Αποστολή στη Λιβύη πρόσφατες αποφάσεις λοιπόν μεταξύ αυτών αποφασίστηκε να ενισχυθεί η αποστολή στα θέματα που ήδη δραστηριοποιείται όπως είναι η καταπολέμηση της παράτυπης μετανάστευσης καθώς επίσης και να ενταθούν οι δράσεις στα πλαίσια της καταπολέμησης της δημοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Ποια ήταν τα αποτελέσματα. Από τότε που συστήθηκε η αποστολή εκπαίδευσε πάνω από 8.000 πρόσωπα σε 360 αποστολές, όπως τεχνικές σύλληψης ε, παράτυπων μεταναστών, ε, ε, διαχείριση χώρων εγκλήματος, διαχείριση στοιχείων σήμασης και συλλογή στοιχείων. Ακόμα και αν δεν είναι το βασικό της μέλημα, έκανε και 61 έργα ε, αξίας περίπου 30 εκατομμυρίων ευρώ. Μεταξύ αυτών ε, βάσεις δεδομένων, ε, ανθρωπίνων δυναμικών, γκαράζ, κινούμενα αστυνομικά τμήματα και άλλα έχει περάσει από την αρχική φάση εκπαίδευσης και κατάρτισης πλέον σε πολύ στοχευμένους τομείς, όπως είναι η σήμανση, η τακτική και τεχνική, ε, αλλά και η συνέχεια που δίνεται, η πλαισίωση και η παροχή συμβουλών. Δηλαδή, τώρα πια η αστυνομία και τα σώματα ασφαλείας του Νίγηρα μπορούν να διαχειριστούν από μόνο τους ε, κάποιες φάσεις κατάρτισης και εκπαίδευση άρα αυτό δείχνει πόσο βιώσιμη είναι η αποστολή εκεί. Επίσης έχουμε και περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα στην Ιαμέη και στο Αγκαντές. Πάντα το κέντρο βάρους στην κατάρτιση και στην παροχή υλικού. Ε, το παράδειγμα του ΑΚΑΤΕΣ λειτουργεί από τον Απρίλιο του 2016 και βεβαίως συμμετέχει σε ε, όλες τις δράσεις και ε, εδρεύει και εκεί κάποιος εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Αποστολής ειδικός για την ανάπτυξη. Ποια είναι τώρα τα μελλοντικά σχέδια και οι προοπτικές και θα τελειώσω εκεί. Ε, στην Άνοιξη θα γίνει μια στρατηγική αναθεώρηση για να προτείνουμε στα κράτη-μέλη μεταξέλιξη και προσαρμογή της αποστολής, υποστήριξη στις αρχές των ήγυρα για να μπορέσουν να αναλάβουν οι ίδιοι την ασφάλεια του πληθυσμού σε όλη την επικράτεια της χώρας. Αυτό θα πρέπει να παραμείνει ε, στον πυρήνα της ε, εντολής της αποστολής. Σε ό,τι αφορά την υποδοχή ε, των μεταναστών, οι δυνάμεις ασφαλείας και ο στρατός έχουν εκπαιδευτεί για το κράτος δικαίου, για το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά αυτό θα εξακολουθήσει να αποτελεί προτεραιότητα για την αποστολή. Και τέλος, τα προβλήματα που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια στον Ήγυρα είναι προβλήματα που γνωρίζουν ε, και άλλες χώρες περιοχής. Άρα θα πρέπει να έχουμε περιφερειακή αντιμετώπιση. Χρειάζεται πρώτα να αναλύσουμε τις ικανότητες ε, για το τι μπορούν να κάνουν οι χώρες G5 ε, σε όλη τη περιφέρεια Σαχέλ, να δούμε τι δυνατότητες έχουν οι ένοπλες δυνάμεις και τα σώματα ασφαλείας των κρατών αυτών για να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ και τώρα θα δώσω το λόγο στον Περιφερειάρχη του Αγκαντές. Κύριε Ανάκο, έχετε το λόγο. Ε, ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, κύριε βουλευτές, είμαι περιφερειάρχης του Ακαδέσ και προσεκλήθηνε εδώ για να καταθέσω τη μαρτυρία μου και να σας πω τι γίνεται τώρα, σήμερα, στο Αγαδές. Ακριβώς όπως είπε και ο προλαλής σας, το Αγαδές, δεν γνωρίζει, είναι ένα μέρος που έχει βορείως την Αλγερία και τη Λιβύη. Με αυτές τις χώρες ε, συνορεύει. Προς Ανατολάς βρίσκεται το Τσάρ και εκεί έχουμε τις περιφέρειες της ε, Ντιφά και άλλη μια περιφέρεια. Εκεί όπου δράει η χαραμστό στο προς έχουμε το Μαλί. Έρημος. Τελείως η περιφέρεια. είναι κάτι σαν μια θάλασσα, όπως την ξέρετε εδώ. Ε, οπότε δεν μπορούμε να έχουμε στεγανή ασφάλεια και ήδη έχουμε 600.000 τετραγωνικά. Είναι η έρημος του Νίγηρα. Οπότε να εξασφαλιστεί η ασφάλεια σε εκείνο το χώρο και σε τόσο μεγάλο χώρο είναι πάρα πολύ δύσκολο. Πάντως η κυβέρνηση έχει βρεθεί σε Ευρωπαϊκή Ένωση ούτω ώστε να αναπτυχθεί η δύναμη αυτή, τη UCAP, ε, από το Μαλί στην περιφερειά μας. Το 2011 η κυρία Μαγερίνη μας επισκέφθηκε και τότε απευθύναμε αυτό το αίτημα γιατί ο κόσμος στον Καντές είπε ναι, ε, μας δίνεται χρήματα Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά θα πρέπει να υπάρχει κάτι συγκεκριμένο. Θα πρέπει να υπάρξει προσέγγιση της Ένωσης με το Αγαδές, γιατί είμαστε πολύ μακριά η περιφερειά μας από τον ΙΑΜΕ την πρωτεύουσα χίλια τόσα χιλιόμετρα από την πρωτεύουσα. Πολλέ φορέ υπάρχουν ρευεργατικέ διαδικασίε στη σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε και έχουμε ζητήσει να υπάρχει κάποιο είδου αντιπροσωπεία τη Ένωση στο Αγαδέ. Ακριβώ διότι η, συγκυρία είναι αυτή που είναι σήμερα από πλευρά ασφαλεία. Το Γιούκα να έρθει. Και αυτό κάτι έκανε. Κάπως ενεργοποίησε τους ε, εταίρους μας γιατί διστάζανε να έρθουν στην περιφέρεια. Μόλις γύρισε σελίδα η κατάσταση με την επανάσταση με τον Καντάφη τους στασιαστές είδατε τι έγινε και στο Μαλία. Οπότε όλοι φοβόντουσαν για τις ομοιρίες. Όλοι φοβούνται την περιοχή μας. Οπότε και είπαμε να έρθει η Γιούκα Ψαχέλ. Αυτό, αυτό θέλαμε. Θέλαμε να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη των εταίρων μας. Αυτό είναι το πρώτο. Αυτή η πρωτοβουλία να έρθει το Γιούκα Ψαχέλ. Δεύτερον, το ucap Ψαχέλ για μας είναι αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην ε, περιφέρεια. Είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση για μας. Οπότε θα πρέπει κάποιος ε, αξιωματός της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ασχοληθεί και με τα οικονομικά να έχει ένα γραφείο που λέμε, λέει ο λόγος στο Γιώκα Ψαχέλ. Άμεση επαφή. Διάλογος. και να έχει κάποια συγγραφή υποχρεώσεων που να είναι πιο ρεαλιστική αυτός ο αξιωματούχος. να έχει συγκεκριμένη αποστολή αυτός ο εκπρόσωπος στα οικονομικά. Τώρα όσον αφορά την ε, αποστολή πολιτικής προστασίας στο ΑΓΑΔΕΣ βεβαίω και υπήρξε ωφέλεια όσον αφορά τις δυνάμεις ασφαλείας. Υπήρξε κατάρτιση, καθημερινή εκπαίδευση, υλικά και το, αυτό, η προμήθεια του υλικού είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι η περιφέρεια θα μπορέσει να προσπαθήσει να αντιμετωπίσει αυτά όλα τα προβλήματα. Το μεταναστευτικό επίσης, πολλές φορές υπάρχουν δυσάρεστες εξελίξεις, οπότε θα πρέπει να έχουν ευαισθητοποιηθεί και οι δυνάμεις ασφαλείας όσον αφορά τη διαχείριση ε, αυτού του προβλήματος, του μεταναστευτικού δηλαδή. Είμαστε ένα σταυροδρόμι. Μεταξύ Μαγρέμπ και Δυτικής Αφρικής. Να, γιατί υπάρχει το μεταναστευτικό. Ε, έχουμε προβλήματα σχετικά σήμερα και οι προερχόμενοι από την Δυτική Αφρική. Από τις χώρες τους έρχονται στο Αγαδές. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι από την Δυτική Αφρική ταξιδεύουν ελεύθερα. Μέχρι το Μανταμά, δηλαδή μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Λιβύη. Όμως, η κυβέρνησή μας για το μεταναστευτικό θέσπισε έναν νόμο για την καταπολέμηση του φαινομένου. Δηλαδή όλοι που έμεσα ή άμεσα εμπλέκονται πρόκειται να υπάγονται σε αυτό το νέο νόμο. Οπότε, οι Αφρικανοί της Δυτικής Αφρικής ε, μεταφέρονται και μεταβαίνουν από το Αγαδέ στη Λιβύη. Κάποτε ήταν τα καραβάνια από Μαλή, από Γκάνα. Συγχρονίστηκαν τα πράγματα. Με τα, με τα 4x4. Οπότε ναι. αυτοί οι μετανάστες από τη Δυτική Αφρική μεταφέρονται, πηγαίνουν στην Λιβύη. Όμως από τότε που έπεσε ο Καντάφη, τότε έχουμε εκεί πέρα μόνο τις στρατοφυλακές. Δεν υπάρχει κράτος στη Λιβύη. Και είναι χωρισμένη η χώρα σε ζώνες επιρροής και τα σύνορα της χώρας με την ε, Λιβύη δεν διέπονται από κάποιους φύλαξη γιατί δεν υπάρχει κράτος στη χώρα. Οπότε στις Φύγανε κανεί στις 6 ώρα, φτάνει το ξημέρωμα στην Λιβύη την επόμενη μέρα, μέσω της ερήμου. Αυτά γινόντουσαν πριν από το 2005, που υπήρχε φυσιολογική ροή μετανάστευσης. Ούτε ο Νίγηρας είχε κάποιο του ειδική νομοθεσία. Από το 2005-2006 μέχρι τώρα είχαμε αυτόν τον νόμο Οπότε φοβούνται αυτοί που έχουν να κάνουν με τους μετανάστες ότι θα συλληφθούν από τις ε, δυνάμεις ασφαλείας. Και έχουν νέους διάβλους, νέες διαδρομές για να παρακάμψουν τις αρχές. Αυτό όμω σημαίνει ότι υπάρχουν κίνδυνοι που ενεδρεύουν. Όπως σας είπα, η έρημος είναι σαν τη θάλασσα. Μπορεί κανείς να χαθεί, μπορεί κανείς να έχει κάποιο πρόβλημα και κανένας δεν πρόκειται να βοηθήσει εάν βρίσκεσαι στην ε, έρημο. Ούτε και κανένας ε, ξέρει το τι έγινε ακριβώς, ποιοι, ποιοι πόσοι πεθαράνε και περνάνε, περνάνε πάρα πολύ καιρός μέχρι να βρουν τις σωρούς. Οπότε ή θα πρέπει να καταστεί νόμιμη αυτή η μετανάστευση και Ευρώπη-Αφρική συνομιλούν από αυτό. Υπάρχει διάλογος για το πώς θα γίνει η διαχείριση της μετανάστευσης. Θα πρέπει να γίνουν οι πρακτικές ρυθμίσεις. Άμα εγώ είμαι από τη Σενεγάλη, από το Μαλί και θέλω ας πούμε να πάω στην Ευρώπη. Θα πρέπει να θεσπιστούν κάποιοι μηχανισμοί ούτως ώστε να μπορεί ένα τέτοιο πρόσωπο να πάει στην Ευρώπη και να μείνει αναγκαστικά. Πάρα πολλοί που έρχονται εδώ αποτελούν, θέλουν να κάνουν κάποια επένδυση στην Αφρική. Οπότε αυτό και ζητούμε ως συνεργασία με την Ευρώπη. Ασφάλεια περισσότερα μέσα για την επίτευξη της ασφάλειας γιατί ο χώρος είναι πολύ εκτεταμένος. Πραγματικά. Ακόμα και τα drones δεν επαρκούν. Τις, εκεί στην Μαντάμα. Και δεν είναι θέμα όπλων. Αυτό λοιπόν και εγώ ζήτησα να απευθύνθηκα στην αποστολή του κάπισα Σαχέλ. στρατιωτική Και το πρόβλημα είναι ότι θα πρέπει να υπάρξει ένα άνοιγμα της υπηρεσίας προς τον κόσμο, γιατί πρόκειται περί πολιτικής, μη στρατιωτικής αποστολής. Το χρειάζεται αυτό ο κόσμος. Και οι πολίτες θα πρέπει να εκπαιδευτούν στα θέματα ασφαλείας. Μόνο έτσι θα ελέγξουμε το χώρο, μόνο αν ο κόσμος είναι στο πλευρό μας πληροφορίες, η διαχείριση του θέματος ασφάλεια. Οπότε έχουμε εκεί και την Περιφερειακή Επιτροπή Ειρήνης. Απαρτίζεται από πολίτες, ξέρουν τα προβλήματα του χώρου. Οπότε υπάρχει και μέθοδος πρόληψης κρίσεων υπήρχε και παρέμβαση όταν η κρίση ήδη είχε ξεσπάσει όπως κάτι πρόβλημα και με του Αρέγ. Και αυτή είναι η προσπάθειά μας να έχει επιχειρησιακό χαρακτήρα αυτή, ε, αυτή η αποστολή όσον αφορά την κοινότητα. να αναβαθμιστεί η Γιούκα Ψαχέλ και να ασχοληθεί και με τους πολίτες, όχι μόνο με τους ε, στρατιώτες. Και έτσι να υπάρχει αναγκαία ευαισθητοποίηση της κοινωνίας για τα θέματα της μετανάστευσης. Είδατε τι γίνεται τώρα στην Λιβύη. Άρα θα πρέπει κανείς να προειδοποιήσει όσον αφορά τους κινδύνους. Και με αυτόν τον νέο νόμο μπορέσαμε να μπλοκάρουμε κάποιους νέους μετανάστες. Έχουν περάσει 5-6 μήνες από τότε που θεσπίστηκε ο νέος νόμος και είπαμε ότι θα πρέπει αυτοί που μεταφέρουν τους μετανάστες να κάνουν κάτι άλλο. Αυτή είναι Άρα με αυτό θα πρέπει να ασχοληθούμε. Θα πρέπει να τους πρόξουμε σε άλλες δραστηριότητε. Μιλάμε για 7.000 περίπου εκεί στην ε, περιοχή μας, στην περιφέρειά μας ε, και επίσης και στην περιοχή που συνορεύει με την Λιβύα. Λιβύη. Να τους πρόξουμε σε άλλες δραστηριότητε για να σταματήσουν να μεταφέρουν τον κόσμο από τη Δυτική Αφρική. 7.000 έχουμε καταγράψει. Τώρα, μια πληροφορία άσχετη με το θέμα της συνάντησης. Άρα έχει σχέση με την ε, διακίνηση προσώπων. Οι διακινητές βρίσκονται παντού. Είναι δίκτυα ολόκληρα. Και από την Δυτική Αφρική, χώρα προέλευσης των μεταναστών, υπάρχουν αυτοί οι διακινητές. που αναλαμβάνουν τις διάφορες φάσεις της διαμετακόμισης. Και υπάρχουν και άλλοι στο Αγαδές, άλλοι στη Λιβύη, άλλοι στην Ευρώπη. Άρα αν θέλει κανείς να καταπολεμήσει αυτή τη λάθρο διακίνηση θα πρέπει να έχει μια σφαιρική, γενική προσέγγιση και όχι μόνο να ασχολείται με τη Σενεγάλη, το Αγαδές ή την Ευρώπη. Και σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Ναι, εμείς ευχαριστούμε κύριε για το πώς ε, μοιραστήκατε αυτές τις ε, πληροφορίες με τρόπο ειλικρινή. Τώρα θα ήθελα να δώσω τον λόγο στον κύριο Άντριου Λέμποβιτς ε, από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Σχέσεων. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και την Υποεπιτροπή που με προσκάλεσε και για την σημασία που αποδίδεται σε αυτό το θέμα. Ελπίζω λοιπόν να σας διαφωτίσει για το ταξίδι σας στον Νίγηρα. Μου ζητήθηκε λοιπόν να κάνω μια παρουσίαση από τη σκοπιά ενός εξωτερικού για τα ζητήματα που αφορούν την Επιτροπή και τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Ήγηρα. Ε, θα ήθελα να τονίσω κάποια πράγματα πριν ξεκινήσω. Δεδομένου του πολύ δύσκολου κλίματος από την Αραβική Άνοιξη, την κατάσταση στη Λιβύη και το μαλη. ο Νίγηρας έχει διάφορες ε, προκλήσεις και η κυβέρνηση τις αντιμετωπίζει εν μέρη με την ε, βοήθεια της διεθνούς ε, κοινότητας ε, και του επαγγελματισμού και της μαχητικότητας των ενόπλων δυνάμεων της χώρας. Θα ήθελα επίσης να τονίσω πως έχω συναντηθεί πολλές φορές με τον παλίστης της αντιπροσωπείας της Ένωσης στον Νίγηρα και πάντα με εντυπωσίαζε η ικανότητά του. Να σας παρουσιάσω πρώτα απ' όλα το πώς ε, έχει λίγο πολύ η χώρα. Από την ανεξαρτησία η χώρα έχει μια πολυτάραχη ιστορία, αλλά με λίγες εξαιρέσεις υπάρχει μια αίσθηση κοινωνικής συνοχής ε, και έτσι δεν υπάρχουν αυτοί οι ενδοκρατικοί πόλεμοι που υπάρχουν παραδείγματος χάρη στο Μαλί και αυτό οφείλεται στο πώς ε, βεβαίως αλληλεπιδρούν οι διάφορες κοινότητες της ε, χώρας αλλά και στις προσπάθειες ε, της ε, κυβέρνησης και διαφόρων φορέων για να διατηρήσουν την ειρήνη. Επίσης η κυβέρνηση έχει καταβάλει μια προσπάθεια από τα δεκαετία του 1990 να αποκεντρώσει εξουσίες και ταυτόχρονα βεβαίως χρησιμοποιεί επιφανείς πολίτες και τις θρησκευτικές αρχές για να μειώσει τις εντάσεις και να διατηρηθεί η ειρήνη. Υπάρχει και η, η πατιαρχή του Νίγηρα για την διατήρηση της ειρήνης και σχετικές αρμοδιότητες ε, του Προέδρου και του Πρωθυπουργού. Ε, είναι ένα σύστημα το οποίο λειτουργεί αλλά δεν είναι τέλειο και πλέον έχει φτάσει στα όρια του. Τούτου λεχθέντος ε, έχει η κυβέρνηση την ευελιξία να αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία ανακύπτουν όπως οι συγκρούσεις μεταξύ των Τούγκου και των ε, διακινητών ε, του ΑΡΕΓ που ξέσπασαν αλλά περιορίστηκαν τελικά. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση και διάφοροι επιφανείς πολίτες ε, μπόρεσαν να προσπάθησαν να ενσωματώσουν διάφορες φυλές, τους του ΑΡΕΓ ιδιαίτερα, πριν από αρκετά χρόνια είχα πάει στην, πρώτη συναυλία στην Νιαμέη ε, μουσικής των Τουαρέγ και αν πάει κανείς τώρα σε γάμο στην Νιαμέη κατά πάσα πιθανότητα η μουσική θα είναι Τουαρέγ αλλά βεβαίως αυτό τα προβλήματα έχουν σχέση με την έλλειψη κράτους ειδικά τη ε, βόρεια της ε, χώρας. Ε, και βέβαια αυτό σημαίνει ότι υφίστανται τεράστια πίεση οι εκπρόσωποι του Βορρά. Ο στρατός παραμένει κυρίως από τις φυλές στην Τζέρμα και Χάουσα στην σύνθεσή του και βεβαίως αγωνίζεται να επιβάλλει την τάξη στον Βορρά και αναγκάζεται να ανέχετε και την διακίνηση από πλευράς αυτών των επιφανών πολιτών και επιχειρηματίων σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες που προσφέρουν στην κυβέρνηση. Επιπλέον, εστιάζουμε πολύ στον Βόρειο Νίγηρα και την περιφέρεια του Αγκαντέζα, αλλά το σύστημα το οποίο περιγράφω δεν μπορεί να αντιμετωπίσει τα ζητήματα σε άλλες περιοχές της ε, χώρας και συχνά ήταν πολύ κατασταλτική η προσέγγιση των αρχών σε άλλες ε, περιοχές. Ε, τα τελευταία χρόνια είχαμε τουλάχιστον 50 επιθέσεις στις δυνάμεις της τάξης από τζιχαντιστές και λοιπούς. Ενώ λοιπόν η κοινωνική συνοχή μπορεί να είναι αποτελεσματική βραχυπρόσφατα, δεν μπορεί να υποκαταστήσει την ύπαρξη κράτους και πρέπει να εστιάσουμε περισσότερο σε αυτά τα τοπικά και εθνικά πολιτικά ζητήματα και να υπάρξει μια πραγματική διακυβέρνηση. Αλλά ταυτόχρονα να είμαστε ξεκάθαροι για το πώς λειτουργεί το κράτος και πώς διατηρεί κάποιες συμμαχίες. Τώρα, κάπως σύντομα, θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα της μετανάστευσης και πώς επηρεάζει κάποια από αυτά τα ζητήματα. Καθώς η μετανάστευση λοιπόν και η λαθροοικονομία ανθούν ε, ε, δεν ε, έδωσαν μόνο δουλειές στον κόσμο στον βορρά της χώρας αλλά δημιούργησαν και κάποια δίκτυα τα οποία βρίσκονταν σε ανταγωνισμό. Όταν υπήρχε άνθηση ας πούμε του κλάδου λειτουργούσαν παράλληλα με χαμηλές εντάσεις, αλλά καθώς ε, οι Τούγκου εξάπλωναν τον τομέα επιρροής τους, άρχισαν κάποιες συγκρούσεις και όταν άρχισε την καταστολή η κυβέρνηση υπό την πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, κάποια από αυτά τα δίκτυα αποδιοργανώθηκαν και έτσι έχασαν το εισόδημά τους ε, και οι λαθροδιακινητές αλλά και οι κοινότητες που εξαρτώνταν από αυτό και δεν είναι μόνο το θέμα του εισόδηματος αλλά το θέμα της δουλειάς ε, και της αξιοπρέπειας ε, που προσπαθούν οι άνθρωποι να έχουν μέσω της δουλειάς δηλαδή πρέπει να θυμόμαστε ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα είναι και το πώς θέλει ο κόσμος να ζήσει, ειδικά οι νέοι της περιοχής. Ενώ η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν επενδύει στο Αγκαντές ε, η βοήθεια αυτή ε, εν ώψη της ε, EUCAP Σαχέλ δεν θα αναπληρώσει το εισόδημα αλλά και την αίσθηση ελευθερίας και ανεξαρτησίας που είχαν οι λαθροδιακινητές. Και βεβαίως υπάρχει και το ζήτημα των σχέσεων μεταξύ των κοινοτήτων και δεν θα μπορέσει η βοήθεια να μπορέσει να προσφέρει κάποια αναλλακτική λύση και απασχόληση για τους διακινητές. Τα λεφτά για τα οποία μιλάμε ε, είναι δεκάδες ίσως εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ στην χώρα και δημιουργούν επίσης ε, έναν κίνδυνο διαφθοράς και σπατάλης ε, στον Βορρά και παραπέρα και βεβαίως ε, είναι μια απτή υπόσχεση, μια υπόσχεση για τον πληθυσμό εκεί, η οποία όμως δεν μπορεί να τηρηθεί και υπάρχουν βεβαίως και τα ζητήματα των προσδοκιών. Και κάτι άλλο το οποίο πρέπει να θυμόμαστε, η μετανάστευση είναι μέρος της ζωής στην περιοχή αυτή και βοηθάει τον κόσμο να επιζήσει σε συνθήκες δύσκολες και οι προσπάθειες να παταχθεί ειδικά εντός ε, της περιοχής ε, του ΕΚΟΒΑΣ ε, διαταράσσουν την κατάσταση εντός και εκτός του Νίγηρα. Οπότε αντιλαμβάνομαι μεν στην Ευρώπη το πολιτικό κλίμα αντιμετώπισης της κρίσης δεν μπορούμε να προσπερνάμε το τι σημαίνει για την περιοχή προσπαθώντας ταυτόχρονα να αντιμετωπίσουμε τις αιτίες. Οπότε το θέμα είναι το τι ε, μπορούν ε, να επιτύχουν ε, οι πολιτικές αυτές. Γιατί η ικανότητα απορρόφησης στον Νίγηρα είναι πολύ χαμηλή και τα προγράμματα αυτά δεν αντιμετωπίζουν τους λόγους για τους οποίους διέρχονται από τον Νίγηρα οι μεταναστές. Δεν διανέμονται παρκώς τα χρήματα και οι άνθρωποι οι οποίοι έκαναν αυτήν την ε, δουλειά θα μπορούσαν να κινηθούν ε, παραδείγματος χάρη στο εμπόριο ναρκωτικών. Και βεβαίως θα επηρεαστεί έτσι και ο κεντρικός και ο νότιος ε, Νίγηρας και θα ε, μπορούσε ίσως να επιδεινωθεί η κρίση της ε, χώρας. Τα δε δίκτυα θα ακολουθήσουν πιο επικίνδυνες ε, διόδους και θα ανταγωνιστούν μεταξύ τους και οι μετανάστες θα κινδυνεύσουν περισσότερο. Η οικοδόμηση αυτή δυνατοτήτων, όπως είπαμε, μπορεί να αντιμετωπίσει κάποια από αυτά τα προβλήματα, αλλά έχει τα όρια της και δεν αντιμετωπίζει ακριβώς τα ζητήματα τα οποία δημιούργησαν αυτές τις καταστάσεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνεισφορά σας και την παρουσίαση αυτή. Είναι αρκετά περίπλοκη η διαδικασία για το ποιο θα πάρει το λόγο. Και από την Ευρώπη και από την Αφρική θα μιλήσουν βουλευτές. Θέλω να σας πω ότι παρευρίσκεται ο πρόεδρος ε, των σχέσεων Ευρωπαϊκής Ένωσης Παναφρικανικού Κοινοβουλίου, κύριος Μιχαήλ Γκάλερ. Θέλετε το λόγο, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Πάρα πολύ εμπεριστατωμένες οι παρουσιάσεις ε, κατατοπιστικές και ενημερωτικές σε ό,τι αφορά την αποστολή μας εκεί, αλλά και αυτά που ακούσαμε από τον κύριο Περιφερειάρχη και τον κύριο Λέμποβιτς. Νομίζω ε, μπορούμε να διδαχθούμε ε, από αυτά που μας λέτε ότι δεν αρκεί να εστιάσουμε στην πόλη του Αγκαντές και να είμαστε παρόντες εκεί. Δεν είναι η μόνη λύση ε, για τα προβλήματα που κρύβονται από πίσω, αλλά μακροπρόθεσμα και ευρύτερα θα πρέπει να ασχοληθούμε με την ευρύτερη περιοχή ακριβώς. Και όλα τα μεμονωμένα μέτρα μπορεί να είναι σωστά από μόνα τους, αλλά αν δεν έχουν συνδυαστεί σε ένα συνολικό πλαίσιο και με μακροχρόνια θεώρηση δεν θα πετύχουν. Θυμάμαι ήδη από το 2011 που υποτίθεται ε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είχε εκπονήσει στρατηγική για το Σαχέλ. Υποθετική λέω, είπε και πραγματική, αλλά το 2011. Και έχουμε την αίσθηση ότι ακόμα είμαστε στα σπάργανα. Βεβαίως δεδομένου και του μεγέθους των προβλημάτων. Άρα, πολιτικά καταρχάς θα έλεγα ότι τώρα αυτό που χρειάζεται δεν είναι ε, μόνο τις παραμονές της Συνόδου Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης, Αφρικανικής Ένωσης, αλλά και στη συνέχεια χρειάζεται ισχυρή δέσμευση ε, των τριών θεσμικών οργάνων και των κρατών μελών για να προχωρήσουμε. Εγώ τώρα μπορεί να κάνω κάποιες μονομένες ερωτήσεις που δεν θα λύσουν το πρόβλημα, το συνολικό. Απλώς επειδή με ενδιαφέρει, κύριε Φερσμέσεν, είπατε ότι στο μεταξύ έχουν ε, αναλάβει την εκπαίδευση των ε, ντόπιων ντόπιοι, εκπαιδευμένοι. Τι γίνεται δηλαδή με τις αστυνομικές δυνάμεις επιτόπου, έχει αλλάξει η συμπεριφορά τους και στην πράξη. Ε, δηλαδή επιχειρησιακά, πώς ε, επεμβαίνουν κατά των διακινητών. Συμβαίνει κάτι τέτοιο με οποιοδήποτε τρόπο. Κάτι που θα μπορούσε να αποτυπώσει κανείς και να διαβάσει και σε αριθμούς ότι κάτι έχει αλλάξει. Καντίστροφα έχω και την ερώτηση προς τον κύριο Ανάκο. Ο λαός στο Αγκαντές. Από τη μια υφίσταται πιέσεις ε, από την κατάσταση αυτή ε, με τις μετακινήσεις. Από την άλλη όμως τους συμφέρει κάποιους γιατί κερδίζουν χρήματα. Δεν ξέρω, πουλάνε τρόφιμα, πουλάνε στέγη, διακινούν, με κάποιο τρόπο βγάζουν λεφτά. ε, δηλαδή ε, υπάρχει ένα ολόκληρο περιβάλλον που δεν έχει καν συμφέρον να αλλάξει τίποτα εκεί. Και αν ενώσουμε τις δυνάμεις μας με την κυβέρνηση της χώρας, μπορούμε να βρούμε εναλλακτική οικονομική δραστηριότητα και να την αναπτύξουμε για το αγκαντές, έτσι ώστε να μην είναι η βασική επαγγελματική δραστηριότητα των κατοίκων και προσοδοφόρα η διακίνηση μεταναστών. Ένα τελευταίο, γιατί πολύ ωραία μας περιγράψατε τα διάφορα δίκτυα και πώς έχουν διεισδύσει τα πλοκάμια τους ε, στην ευρύτερη περιοχή, που είναι η μεγάλη υπάρχει δυνατότητα να κάνουμε κάτι στις χώρες προέλευσης τους, πατρίδες τους, πριν φτάσουν στο Αγκαντές, να συνεργαστούμε κάπως με τις αρχές, έτσι ώστε και εκείνοι να έχουν συμφέρον να σταματήσουν τους διακινητές. Κάποτε είχαμε ένα συνάδελφο που μου είπε, μία από αυτές τις χώρες, ήταν η πατρίδα του, ότι το πρόβλημα ποιο είναι. Όταν μαζεύουν τα χρήματα οι διακινητές από τους μετανάστες, Το πρώτο που κάνουν είναι να λαδώσουν τις τοπικές αρχές. Μήπως να το πάρουμε αλλιώς. Ένας ε, υπάλληλος ε, κρατικών αρχών που συλλαμβάνει ένα διακινητή να αμείβεται. Γελάει η κυρία Λόζινγκ. Μα τι με τους διακινητές είσαστε, γιατί γελάτε. Θα πρέπει να καταλάβετε πώς έχει κατάσταση επιτόπου. Έχουν συμφέρον οι άνθρωποι να γίνει κάτι τέτοιο. Και αν εγώ είμαι αστυνομικό, ξέρω εγώ είμαι υπάλληλο και ε, δωροδοκούμε και χρηματίζομαι από τον διακινητή, είναι διαφορετικό από το να έχω ανταμοιβή. Ε, όταν συλλαμβάνω ένα διακινητή. Δηλαδή καλύτερα να γίνεται νόμιμο μια επιβράβευση παρά να αλλαδώνεται παράνομα. Δεν ξέρω αν είναι αυτό ρεαλιστικό. Σίγουρα θα έχουμε περισσότερες ερωτήσεις παρά απαντήσεις αλλά μου Ευχαριστώ. Thank you very much. Ε, ευχαριστώ πολύ. Και τώρα θα ήθελα να δώσω λόγο ε, στους συναδέλφους από την Αφρική. Ζητώ συγγνώμη αν κάνω λάθος στην προφορά των ονομάτων σας. Ο γερουσιαστής Γκομέρ ε, απουσιάζει, οπότε θα δώσω πρώτα το λόγο στο γερουσιαστή Βακύρη. Ζητώ συγγνώμη για τα ονόματα. Δεν ξέρω και τα μικρά σας. Θα μπορούσατε να συστηθείτε παρακαλώ. Έχετε το λόγο. Uh, thank you, Mrs. Chair. Ευχαριστώ, Ε, είμαι ο Μαλέ ο Οικίλη από την Γερουσία της ε, χώρας ε, του Μαλή της Νιγηρίας με συγχωρείτε ειδικά χαίρομαι που μπορώ να μιλήσω σήμερα για την τρομοκρατία καθώς αντιμετωπίζουμε εμείς τον Μπόκο Χαράμ απαγωγές, εμπόριο όπλων ε, λάθρο διακίνηση ανθρώπων κτλ. Η Νιγηρία είναι η πολυπληθέστερη χώρα της Αφρικής. Είναι μια περιφερειακή δύναμη στην Δυτική Αφρική και βεβαίω οτιδήποτε συμβαίνει στην Νιγηρία ενδιαφέρει όχι μόνο τη Δυτική Αφρική και την Αφρική αλλά όλους μας γιατί το πρόβλημα το οποίο θα δημιουργηθεί θα είναι πάρα πολύ μεγάλο για να το διαχειριστούν οι χώρες. Έχουμε τα εσωτερικά μας προβλήματα που σχετίζονται με το διεθνές έγκλημα. Έχουμε και το IPOB κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ζητάνε ανεξαρτησία από την γενία και συχνά καταφεύγουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί έχουν διπλή υπηκότητα και έχουμε προβλήματα στο να δικαστούν κτλ. Ε, δεν τους εκδίδουν τα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε το θέμα του Μπόκο Χαράμ, το οποίο δεν είναι Ισλαμικό, ε, γιατί όπως ξέρετε το Ισλάμ σημαίνει ειρήνη. Και από τα ευρήματα τα οποία έχουμε, αποτελούνται από ανθρώπους από διάφορες εθνικότητες, όχι μόνο Νιγηριανούς, από τις περιοχές ε, της ε, Δυτικής Αφρικής και παραπέρα. Συνελήφθη μάλιστα και ένας Ευρωπαίος υπήκος ε, μεταξύ των μαχητών. Δεν είναι λοιπόν θέμα θρησκείας. Απαγωγές επίσης πάρα πολλές. Ε, έχουμε και θύματα. Ως ε, κοινοβούλιο η Εθνοσυνέλευσή μας έχει περάσει ένα νόμο που τιμωρεί με θάνατο την απαγωγή. Ανεξαρτήτως αν το θύμα πεθάνει ή όχι, γιατί υπάρχει ε, αυτή η πιθανότητα. Έχουμε επίσης ε, παράνομα όπλα που μπαίνουν στη χώρα, κάποια από αυτά από την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάποια από αυτά από δυνητικά μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έχουμε σταματήσει κοντέινερ ε, όπλων από υποψήφιες χώρες, αλλά από το Ιράν και από αλλού. Προσπαθώ να σας περιγράψω δηλαδή το τι συμβαίνει με το οργανωμένο έγκλημα στην Ιγυρία. Η Ιγυρία ε, Έχει μια. Θα τη χαρακτηρίζα ως μια μεγάλη αδελφότητα και συνδέονται και οι άλλες χώρες με την οικονομία μας. Έχουμε την ε, λεγόμενη συνθήκη Έκοβας ε, της Δυτικής Αφρικής που προβλέπει ελευθεριακή διακίνηση αγαθών και υπηρεσιών και πρόσβαση στις αγορές και καμιά φορά τα αγαθά τα οποία έρχονται στην χώρα μας ε, έρχονται μέσω γειτονικών χωρών και μέσω λαθρεμπορίου. Και Βεβαίω υπάρχει και η απειλή για τους γειτονές μας όσο επιτρέπουν ε, να διοχετεύονται μέσω των χωρών τους ε, όπλα και τέτοια πράγματα. Καθίσαμε λοιπόν να δούμε ως νομοθέτες ε, το τι συμβαίνει. Επίσης ε, ε, αντιμετωπίζουμε και το κυβερνό έγκλημα, την περίφημη Νιγηριανή απάτη και αυτό το ποινικοποιήσαμε. Έχουμε επίσης τον νόμο περί ξεπλήματος χρήματος και τρομοκρατίας που περάσαμε πριν από δύο χρόνια για να αντιμετωπίσουμε ακριβώς το θέμα του ξεπλήματος χρήματος και των σχετικών αδικημάτων. Τι συμβαίνει όμως λοιπόν. Ο πρόεδρός μας έχει πάει σε άλλες χώρες της ε, περιοχής για το ζητήματα της ε, τρομοκρατίας και για να το αντιμετωπίσουμε αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε την διαφθορά. Για να σταματήσει αυτό ε, θα πρέπει να μας βοηθήσετε εσείς που λαμβάνετε τα λεφτά των διεφθαρμένων. Δεν θα αναφέρω λοιπόν κάποια χώρα συγκεκριμένη. Ας δούμε τι γίνεται παραδείγματο χάρη με τον νόμο περί κληρονομιάς. Ε, μπορούν να έρχονται οι Νιγηριανοί σε μια συγκεκριμένη χώρα της Ένωσης να αγοράζουν ακίνητα, να τα κληροδοτήσουν και δεν χρειάζεται καν να, να γνωρίζουν το κράτος ποιος είναι ο ιδιοκτήτης αρκεί να πληρώνει το φόρο κληρονομιάς. Ε, πρέπει να επαναπατριστούν τα χρήματά μας λοιπόν, τα οποία με, με διαφθορά έρχονται στις ε, χώρες σας. Και έχουμε και τις ε, πολυεθνικές που διαχειρίζονται οι πολίτες σας. Για το Μποκοχαράμ. Έχουμε μια πολυεθνική δύναμη με έδρα το Τσάντ, αλλά εξακολουθούμε να έχουμε κάποια προβλήματα όσον αφορά την συνεργασία. Ε, οι δυνάμεις αυτές ήταν αγγλόφωνες, ε, γύρω-γύρω υπήρχαν γαλλόφωνοι πληθυσμοί, υπήρχε και αυτό το ζήτημα. Για την κοινωνικο-οικονομική βάση του Νιγηριανού κράτους, η οποία ε, πράγματι δημιουργεί αυτά τα ζητήματα ριζοσπαστικοποίησης κτλ. Τι τους κατοίκους του Δέλτα του Νίγηρα που αισθάνονται ότι υφίστανται μόνο εκμετάλλευση και δεν εκμεταλλεύονται τον πλούτο κτλ. Ο πρόεδρος έχει νομοθετήσει σχετικά και θα αντιμετωπιστούν τα προβλήματα από το 2020 και μετά θα έχουν αντιμετωπιστεί όλα. Λοιπόν, μετά έχουμε και την Επιτροπή Αναπτύξεως ε, του Βορρά που θα ασχοληθεί με την ανοικοδόμηση και ένταξη και όλα τα σχετικά ζητήματα της ε, περιοχής εκεί γιατί υπάρχουν πολλά ορυκτά και άλλα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να επέλθει η ειρήνη και να μην ε, μπαίνει ο κόσμος σε συμμορίες για τη διαχείριση των συνόρων Μέσω του ΕΚΟΒΑΣ έχουμε την συνεργασία των αρχηγών των υπηρεσιών ασφαλείας, αστυνομίας και λοιπόν, για να μοιραστούν ακριβώ τις πληροφορίες ε, που αφορούν τα σύνορα. Τι θέλουμε εμείς από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, δεν θέλουμε βοήθεια, βοήθεια, βοήθεια. Όχι. Ε, πρέπει να μας βοηθήσετε εκεί που έχουμε προβλήματα ε, να τα αντιμετωπίσουμε, να δημιουργηθούν δυνατότητες, να υπάρχει πρόσβαση σε εξοπλισμό. Έχουμε αλφατζετ, τα οποία αγοράσαμε από τη Γαλλία και είναι πάρα πολύ δύσκολο. Ε, βλέπουμε ότι πλέον είναι απερχαιωμένα αεροσκάφη και δεν ε, έχουμε πια ανταλλακτικά. Ούτε νέα παράγονται βεβαίως. Οπότε πρέπει να μας βοηθήσετε για να πολεμήσουμε ακριβώς του τρομοκράτε πρέπει να μα βοηθήσετε και στην πλευρά του εξοπλισμού, των πληροφοριών, εκπαίδευση του προσωπικού κτλ. Για το θέμα της ε, λαθροδιακίνησης. Χτες, εδώ νομίζω στην ίδια αίθουσα όπου ακούστηκε ότι χάνονται δισεκατομμύρια λόγω αυτού του ζητήματος, ειδικά στην Ιταλία, όπου είναι κυρίως ε, συμμορίες ε, Νιγηριανών και, με και κορίτσια από την Νιγηρία τα οποία τα εκμεταλλεύονται. Το ερώτημα είναι πώς τους τιμωρείτε. Γιατί αν τους ε, εκμεταλλεύονται, αν υπάρχουν προαγωγή, δεν μπορεί να τιμωρείται μόνο τα κορίτσια και όχι αυτούς που τους εκμεταλλεύονται. Δεν ξέρω αν και ο συνάδελφός μου έχει να πει κάτι. Ο Μοχαμενταλή εδώ ο συνάδελφος. Σας ευχαριστώ. Θα λέει πρώτος. θα δώσουμε τον λόγο με την σειρά στους ευρωβουλευτές ε, και στους βουλευτές ε, του Αφρικανικού Κοινοβουλίου και των Αφρικανικών Κοινοβουλίων. Τώρα, επόμενος συντονιστή. είναι η κυρία Λέζινγκ. Έχετε τον λόγο. <clears throat> Ευχαριστώ πολύ. Θα προσπαθήσω λίγο στα σχόλιά μου να συμπεριλάβω και αυτά που ακούσαμε χτες. Περιμένω λίγο να βάλουν ακουστικά. Ωραία. Στα σχόλιά μου έλεγα θα ήθελα να συμπεριλάβω αυτά που ακούσαμε χτες για την κατάσταση στο Μάλι. Και θα όσα ακούσαμε σήμερα. Οφείλω να πω το εξή απλούστατα, ότι σιγά σιγά ή όλο και περισσότερο αναρωτιέμαι τι κάνουμε εμείς Ευρωπαίοι πολιτικοί. Έχω την αίσθηση ότι κόβουμε ένα κεφάλι της Λερναίας Ήδρας και μετά βγαίνουν 10 και 100 καινούργια κεφάλια επικίνδυνα αξιολογούμε την πολιτική του Καντάφη και τα λοιπά. Και πού καταλήγουμε. Φαίνεται από τη συζήτηση ότι αυτό ήταν πραγματικά το ένα κεφάλι της νέας ίδρας που καταληγουμε φαινεται απο τη συζητηση οτι αυτο ηταν πραγματικα το ενα κεφαλι της νεας που κοψαμε και έπονται περισσότερο. Ακούσαμε ότι η μετανάστευση περνάει από την έρημο, η οποία έρημος είναι σαν μια μεγάλη θάλασσα. Και ακούσαμε επίσης ότι οι άνθρωποι αυτοί σε αυτή την έρημο, τη θάλασσα της έρημου, χάνουν τη ζωή τους. Και ερχόμαστε να χειροκροτήσουμε τα αποτελέσματα της περιχαράκωσης στη Μεσόγειο, ότι ο κόσμος σταμάτησε να πνίγεται. Ωραία, δεν πνίγεται, ε, πεθαίνει στην έρημο τώρα. Έχω την αίσθηση ότι χτίζουμε τείχη γύρω-γύρω, στέλνουμε όπλα, ε, εκπονούμε συστήματα φύλαξη στο σύνορο. Τι γίνεται, γίνονται όλο και πιο χοντρά τα τείχη και από πάνω βάζουμε και καπάκι. Αυτό το ξέρει η κάθε νοικοκυρά που μαγειρεύει, όταν ε, κάνει τέτοια πράγματα και τα καπακώνει και όλες, κάποια στιγμή θα εκραγεί αυτή η χύτρα. Χρειάζεται ανάλυση των συγκρούσεων εκεί και κάποια στιγμή να έχουμε μια στρατηγική. Μια οποιαδήποτε στρατηγική που να περιλαμβάνει κάτι διαφορετικό από την απόκρουση της μετανάστευσης. Και πραγματικά ρωτιέμαι εδώ πέρα. Ακούω συνέχεια για παράτυπη μετανάστευση, μετά παράνομη μετανάστευση, μετά λάθρο μετανάστευση. Μετά λέει φροντίζουμε να διαφυλάσσονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Οι άνθρωποι έχουν δικαίωμα στο άσυλο. Και ποιος ε, αξιολογεί τι εστί νόμιμη και τι παράνομη μετανάστευση. Μα η μετανάστευση εκεί στην περιοχή ακούσαμε ότι είναι φυσιολογικό. Και έχουμε στρατιώτες που τους πληρώνουμε εμείς και πυροβολούν μετανάστες. Πρώτα πυροβολούν, τους σκοτώνουν και μετά ψάχνουν αν ήταν νόμιμος μετανάστης ή παράτυπος ή αν έχει στη τσέπη του αίτηση ασύλου ή απλώς ήταν ένας έμπορος πλανόδιος ε, στην έρημο. Αυτά είναι σημεία μεμονωμένα από τις δικές σας τοποθετήσεις. Εχθές, για παράδειγμα, από εξέχοντα μέλη του πάνελ και ικανότατα ακούσαμε ότι φοβόμαστε μήπως το Μαλί εξελιχθεί σε νέο Αφγανιστάν. Εγώ θα το επεκτείνω σε ολόκληρη τη Βόρεια Αφρική, τη Βόρεια περιοχή της Αφρικής, μήπως γίνει ολόκληρη ένα Αφγανιστάν. Στο παρελθόν υπήρχαν εύκολοι δρόμοι να πάει κανείς από τη Δυτική Αφρική ε, μέσω της Μεσογείου δεν είχαμε μαζικού θανάτου στην έρημο. Αυτά προέκυψαν αφότου η Frontex περίπολη ε, στην Αφρικανική ακτή πάνω κάτω. Και να μην ξεχνάμε ότι για όλες αυτές τις αποστολές χρησιμοποιούνται κονδύλια από την αναπτυξιακή βοήθεια. Αυτό το λέω για τους συναδέλφους μας από την Αφρική. Εσείς αυτό πώς το βλέπετε. Από τη μια λέμε ότι θέλουμε να καταπολεμήσουμε τις αιτίες της φυγής και παίρνουμε λεφτά από την διευκόλυνση για την ειρήνη που είναι αναπτυξιακή βοήθεια και τα πάμε σε στρατιωτικές ικανότητες όλο και περισσότερο. Τι θα πει καταπολέμηση των αιτίων της φυγής. Δεν τα προλαβαίνω να σας τα ε, κατονομάσω όλα και να τα απαριθμίσω. Κάτι θετικό να πω. Αυτό το συμβούλιο, το ερνευτικό και τη δουλειά που κάνει, πραγματικά θέλω να την εκθίασω. Είναι το μοναδικό και το πρώτο που ακούω που αξίζει να υποστηριχθεί. Αξίζει να υποστηριχθεί. Αν εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση ε, κάπου μπορούμε να λύνουμε ε, ειρηνικά τις σειράξεις και πώς μπορεί να γίνει πρόληψη και ειρηνική διευθέτηση των συγκρούσεων. Και χρειαζόμαστε μια συνολική στρατηγική. Και κύριε Γκάλερ, δυστυχώς ε, πρέπει να επανέλθω σε αυτό που είπατε εσείς όταν γέλασα προηγουμένως. Πραγματικά ήμουν υποχρεωμένη, δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Αυτό μας έλειπα. Βάλουμε και λίτρα τώρα. Θα τους επικηρύξουμε τους διακινητές. Αυτό είναι άλλη μια βεβαιασμένη και απελπισμένη κίνηση ε, σε αυτό το τοίχο που χτίζουμε. Κάποια στιγμή αυτή η χύτρα που την έχουμε κλείσει γύρω-γύρω και βάλει και καπάκι από πάνω θα εκραγεί. Ανησυχώ. Εγώ δεν ανησυχώ για τις μεταναστευτικές ροές. Αλλά θα πρέπει να σκεφτούμε πώς θα τις ε, διοχετεύσουμε στην νόμιμη μετανάστευση. Αυτό για το οποίο ανησυχώ είναι τι θα γίνει με αυτή τη χύτρα που κοχλάζει τώρα και είναι γεμάτος ατμός εκεί το καζάνι αυτό. Όταν σκάσει, τι θα γίνει όταν εκραγεί. Ευχαριστώ πολύ. Ο αξιότιμος κύριος Μοχάμετ Άλλη από την Ιγυρία. Thank Ευχαριστώ πολύ. Καλά το είπατε, Μοχάμετ Άλλη Ντίλ. Είμαι από την ε, Νιγηρία. Να μιλήσουμε για το θέμα μας, δηλαδή το πώς θα αναβαθμίσουμε τις δυνατότητές μας για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Και βέβαια το θέμα αφορά και τον Ήγερα και άλλες αφρικανικές χώρες, όπως είπε ο συνάδελφος, είναι ενδυμικά τα φαινόμενα της ε, τρομοκρατίας και είναι κάτι το οποίο έχει πλήξει όλο τον κόσμο. Επομένως, θα πρέπει να το καταπολεμήσουμε. Ο Μπουχάρη, ο πρόεδρος Τι έκανε το 2015. Μετακόμισε τις ε, βάσεις των ενόπλων δυνάμεων της χώρας ούτως ώστε να είναι πιο κοντά στις περιοχές που υπήρχε τρομοκρατία να την καταπολεμήσει. Να έχει την έδρα του στρατό και το ε, επιτελείο τέλο πάντων εκεί όπου υπήρχε το πρόβλημα με αυτή την μετακίνηση είχαμε καλύτερες επιδόσεις στο θέμα της ασφαλείας και κάτω τη της τρομοκρατίας. Τσάντ, Νίγηρα και Καμερούν. Αυτές τις τρεις χώρες ε, πρέπει να επισκεφθεί κανείς όπως και έχει γίνει για να δει τι γίνεται γιατί θα πρέπει εκεί να υπάρξει συνεργασία κατά της τρομοκρατίας. Έτσι και τα καταφέραμε καλύτερα για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας. Και για το οργανωμένο έγκλημα μίλησαν οι συνάδελφοι. Διότι αφορά ακριβώ και άλλες χώρες το φαινόμενο. να δούμε τι έχει γίνει. Χρειάζεται συνεργασία που έγινε και με την Ισπανία. Να δούμε επομένως ποιο είναι το κόστος του φαινομένου επίσης. Ε, προς τούτο θα πρέπει να υπάρξει συνεργασία. θα πρέπει να τα δούμε. Έχουμε αυτού τους 26 που σκοτώθηκαν. Θα πρέπει να γίνει η έρευνα, η νεκροψία. Αλλά από τι πέθαναν. θα τον περιοριστώ στο θέμα μας. Πώς δηλαδή θα περιορίσουμε την έκταση του φαινομένου και του εγκλήματος της τρομοκρατίας. και η σημερινή κυβέρνηση της χώρας μας έχει υποσχεθεί ότι θα καταπολεμήσει την τρομοκρατία και από το IPA, ένα πανεπιστήμιο, έχει ε, αναγνωριστεί η προσπάθειά της και οι επιδόσεις της. Όσον αφορά δηλαδή το να πώς θα μειωθούν τα θύματα της τρομοκρατίας. και πρόκειται για μια μάστιγα που εξαπλώνονται στην Αφρική. Και αντίθεμα ότι είπα εμείς, συμβάλλουμε πολλούς τρόπους και δεν είναι θέμα όλων αυτών των χρημάτων που φύγανε από την χώρα και από την Ήπειρο. θέμα ε, του επαναπατρισμού, του τι γίνεται με τις τράπεζες. Ε, αυτό είναι το πρόβλημα για πολλούς όμως και αυτά θα πρέπει να δούμε. Αυτά τα προβλήματα. Τα όπλα που χρησιμοποιούνται. Τα όπλα φτιάχνονται στην Ευρώπη και αλλού και έρχονται στην Αφρική ούτω ώστε οι Αφρικανοί να πολεμάμε ένα στον άλλο. Οπότε καταπολεμάται η, η τρομοκρατία, αλλά τι θα γίνει το πρόβλημα των όπλων που λαθρέα μπαίνουν στη χώρα. Όπλα που κυρίως προέρχονται από χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως είπε και ο συνάδελφος. Χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μικρά όπλα. Θα φέρνουν για τους εγκληματίες και τους τρομοκράτες. Α, είναι το, το πρόβλημα ότι διακυβεύεται και η δική σας ασφάλεια. με γίνεται στην Αγγλία και τελικά τα όπλα που χρησιμοποιούνται φτιάχνονται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως και τα πυρομαχικά Άρα όλοι θα πρέπει να θεωρήσουμε ότι είμαστε μαζί σε αυτή την προσπάθεια και να επιληθεί αυτό το πρόβλημα της λαθρεμπορίας όπλων προς την Αφρική. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Κυρία Άννα για τους σοσιαλιστές έχει το λόγο. Ευχαριστώ εγώ. Πολύ σημαντικά αυτά που είπαν οι συνάδελφοι από το Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστούμε και τους προσκεκλημένους μας και κυρίως τον κύριο Ανάκο που ξεκάθαρα μας τα εξήγησε. ότι η έρευνα μεταξύ Νιγηρίας και Νίγηρα και Λιβύης είναι ο τόπος για όλους αυτούς τους μετανάστες που για να διέλθουν είπαμε τι γίνεται με αυτούς που πνίγονται στην Μεσόγειο και ανακαλύπτονται τα πτώματά τους χρόνια μετά οπότε είναι πάρα πολλοί όσοι είναι θύματα αυτής της λαθροδιακίνησης. Επίσης, μας εξηγήσατε ότι δεν έχουν να κάνουν τίποτα άλλο οι νέοι στην περιοχή σας, οπότε αυτό που κάνουν είναι να γίνονται λαθροδιακινητές. παράνομη δραστηριότητα αλλά και περισσότερος ο κίνδυνος για τους ε, μετανάστες και όμως έχουν τις περισσότερη δουλειά οι λαθροδιακινητές γιατί είναι χαζή η πολιτική μας το ότι δεν έχουμε βρει κάποιους νόμιμους ε, τρόπους ε, ελέγχου της μετανάστευσης η Επιτροπή, το Συμβούλιο, οι χώρες μας θα πρέπει να μην αγνοούν την πραγματικότητα να μην διαφορούν για την πραγματικότητα, να βρεθούν ε, νόμιμοι τρόποι. Είναι γελίος θεσμός η μπλε κάρτα που χρησιμοποιεί πάσα Ευρωπαϊκή Πρεσβεία. Να βρεθεί νόμιμος τρόπος για όσους θέλουν να έρθουν στην Ευρώπη. Να ζητήσουν ε, άσυλο, να φύγουν από την καταπίεση, την καταστολή, τη δίωξη. ακόμα και οικονομικοί μετανάστες, δεν έχουν άλλο τρόπο παρά μόνο να εμπιστευτούν τους διακινητές. Άρα εμείς δημιουργούμε δουλειά για αυτούς. Ακριβώς όπως είπε ο κύριος Ανάκο και ο κύριος ε, Λέμποβιτς. Και βέβαια οι διακινητές έχουν σχέση και με δίκτυα εγκληματιών και στην Ευρώπη και παντού. Και τελικά χρηματοδοτείται η τρομοκρατία. Λάθρο εμπόριο τσιγάρων, όπλων κλπ. Τα ξέρουμε καλά. Από την Μπόκο Χαράμ οργανώσεις σε όλο το Σαχέλ και στην Ευρώπη. Τα ξέρουμε το πόσο ασχολείται η μαφία με τέτοιε δραστηριότητε. Έχει στη Λιβύη, είναι business, τρομερή αυτό. Επομένω εμείς, εμείς φταίμε και οι κυβερνήσει μα με το να αγνοούν την πραγματικότητα. Και το να πληρώνουμε τις στρατοφυλακές δεν είναι λύση αυτή, είδαμε τι έγινε. Κοροϊδεύουμε τους εαυτούς μας, κάνοντας και προσποιούμενοι ότι έχει υπάρχει κράτος στη Λιβύη. Και βέβαια δεν το λέω από νοσταλγία για τον Καντάφη που ήταν μέγας καταπιεστής. Τα έχω δει με τα μάτια μου. Η πτώση του καθεστώτος Καντάφη δεν ήταν από τα έξω επέμβαση. Ήταν ο λαός που ξεσηκώθηκε. βιασμό της βάρος της Ευρώπης. Οπότε θα πρέπει τώρα να σταματήσουμε να βοηθάμε τους διακινητές και το πόσο έντονη δραστηριότητα έχουν και έτσι να καταπολεμήσουμε και τα εγκληματικά δίκτυα. Εσείς να τα πείτε από την ε, Παναφρικανική Ένωση. Πέστε τα όταν γίνει η συνάντηση κορυφή με την Ένωση. Να τους τα πείτε. Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Και βέβαια όσον αφορά την ασφάλεια οι συνέπειες είναι τρομερές. Πρόθυμο μπορεί των μικρών όπλων όπως τα είπατε συνάδελφοι. το 2008 επί Γαλλικής Προεδρίας υιοθετήσαμε εκείνη την κοινή θέση ε, κατάληξαμε σε δέσμευση των κρατών μελών για να σταματήσει ακριβώς αυτό το λαθρεμπόριο από την Ευρώπη προς την Αφρική και προς όλο τον κόσμο και τα όπλα μαζικής καταστροφής και την πρόσφατη έκθεση έχουμε που καταγγέλει ότι τα περισσότερα κράτη δεν σέβονται την δεσμευσή τους. Και εσείς κύριε Γουακίλη, έχετε όλα τα δίκαια του κόσμου. Όχι, δεν είναι θέμα βοήθειας και ενίσχυση προς την Αφρική. Όλα αυτά είναι διασπάθηση των χρημάτων των Ευρωπαίων φορολογουμένων. Το πηγάδι δίχως πάτο. Ε, θα πρέπει λοιπόν τα χρήματα να πιάσουν τόπο βοηθώντας την κοινωνία εκείνους που ε, λογοδοτούν στις κυβερνήσεις τους στην Αφρική. Να σταματήσει υποστήριξη προς την κλεπτοκρατία και τις διεφθαρμένες κυβερνήσεις. Α, είχαμε τα Panama Papers, τώρα τα Paradise Papers και βγήκαν στο φως όλα αυτά. Τι γίνεται με την κλεπτοκρατία. Και το σύστημα στην Ευρώπη που οδηγεί στο ξέπλυμα χρήματος και που τελικά τα χρήματα τέτοιων δραστηριοτήτων από την Αφρική κατελήγουν σε επενδύσεις στην Ευρώπη και το 2013 επίσης είχε ασχοληθεί με το πρόβλημα Επιτροπή Ανάπτυξης. Λέγαμε για την Αραβική Άνοιξη, αλλά τελικά το θέμα ήταν γενικότερο. Το πώς η Ένωση και η Κομισιόν ε, ασχολήθηκαν με ακριβώς την επιστροφή κάποιων κεφαλαίων στις χώρες προέλευσης. Ναι, αυτά θα πρέπει να γίνουν. Αυτό χρειάζεστε και αυτό χρειαζόμαστε και εμείς. Αλλά θα πρέπει οι κυβερνήσει μα να ακούσουν πραγματικότητα. Κάποιο να του την εξηγήσει. Γιατί αυτό να το κάνουν οι Αφρικανικέ χώρε, η Αφρικανική Ένωση που πολλέ φορέ σιωπά. Υπάρχει συνενοχή με την κλεπτοκρατία στην Αφρική. Για δικό μας πρόβλημα και άρα όλα αυτά θα πρέπει να τα ακούσουν οι κυβερνήσεις. Θα είναι μεγάλη ευκαιρία συνάντηση κορυφή Ευρώπη Αφρική και για την μετανάστευση που θα πρέπει να τύχει διαχείριση και να υπάρχουν ασφαλείς τρόποι διαχείρισης, ε, νόμιμοι τρόποι και να κόψουμε τη δουλειά των δικτύων και των διακινητών. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Ο επόμενος. Α, μια ε, ε, τελική, τελευταία ερώτηση προς τους φίλους από την Αφρική. Α, συνεχίζουμε να υποκρινόμαστε ότι ασχολούμαστε με το πρόβλημα και ότι κάτι κάνουμε γι' αυτό όταν αγνοούμε, κάνουμε ότι υπάρχει κράτος στη Λιβύη και έχουμε αυτόν τον πόλεμο δι' που γίνεται εκεί κάτω, στη Σαουδική Αραβία, στη Λιβύη. με τους σαλαφιστές, με τους εξτρεμιστές, με τη στατολόγηση τρομοκρατών από αυτά τα καθεστώτα και να λέμε ότι υπάρχει αναγνωρισμένη κυβέρνηση στη Λιβύη, αναγνωρισμένη από τον ΟΗΕ, που δεν μπορεί να ελέγξει τίποτα. Μα είναι δυνατόν και εμείς, αλλά και η Αφρικανική Ένωση, να φοβόμαστε, να παραδεχτούμε ότι υπάρχει και ένα τεράστιο κενό διακυβέρνησης να συνεργαστούμε και να σταματήσουν οι αυταπάτες αυτές και η υποκρισία. Και εκπαιδεύουμε και την ακτοφυλακή. Μα όχι, δεν κάνουμε αυτό. Πληρώνουμε τις πολιτοφυλακές. Είμαστε συνένοχοι με τα αποτρόπια αυτά τα εγκλήματα που κάνουν αυτοί. Σας ευχαριστούμε πολύ, λέει Πρόεδρος. Έχουμε δύο μελετές ακόμα. Και μετά θα ήθελα να δώσω το λόγο στα μέλη του πάνελ για να απαντήσουν. Γιατί έχουν καταφτάσει και τα μέλη του πάνελ για το επόμενο θέμα μας, που είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό για το Ιράκ. Και τώρα το λόγο έχει η κυρία Αϊχάτα Χαϊτάρα από την ομάδα των γυναικών ε, στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Εξ ονόματος του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανητές του φόρουμ αυτού μεταξύ των δύο κοινοβουλίων μας γιατί πραγματικά πολύ καιρό περιμέναμε αυτή τη συνεργασία. Η στρατιωτική επέμβαση στη Λιβύη ε, πυροδότησε άνευ προηγουμένου έκρηξη στην Αφρική γενικότερα και ειδικότερα στο Σαχέλ. Θα πρέπει οι βουλευτές να ασχοληθούν έτσι ώστε η διεθνής δικαιοσύνη ε, να ε, τιμωρήσει τους ενόχους. Και μιλώ για το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο. Δεν μπορούμε να έχουμε δικαιοσύνη δύο ταχυτήτων μόνο Αφρικανούς παραπέμπουμε ε, στο δικαστήριο. Μέγας λόγος γίνεται για τη Λιβύη, αλλά όχι πολύ μεγάλος για τις ε, αιτίες. Το είπε ο πρόεδρος του Κοινοβουλίου μας. Θέλω να το επαναλάβω κι εγώ. Ε, εγώ κατάγομαι από το Μαλί και ζω στο βορρά της χώρας και καθημερινά στο πετσί μου τι συμβαίνει. Υπάρχει τεράστια ανασφάλεια παγκοσμίω και ιδιαίτερα στην Αφρική. Επίσης σε κάποιες αφρικανικές χώρες γίνεται κακή διαχείριση των εκλογών και αυτό οδηγεί σε σειράξεις μικρότερες μένα, αλλά μπορεί να φτάσει αυτό μέχρι εμφύλιο πόλεμο ε, μεταξύ διαφόρων πολιτικών παρατάξεων και κομμάτων. Θα έλεγα λοιπόν ότι η ανάμεξη στα εσωτερικά ε, των αφρικανικών χωρών θα πρέπει να σταματήσει ε, από πλευράς δυτικών κρατών, τουλάχιστον να μετριαστεί και να γίνει πιο δίκαιη. Είναι πολύ ε, σημαντική η συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι' αυτό θα πρέπει να έχουμε σχέσεις αμοιβαίως αμοιβαίως-εποφελείς και όχι η κατάσταση οι ε, σχέσεις προϊσταμένου υφισταμένου ή μεγάλη χώρα προς μικρή. Το 2013 υπήρξε σύνοδος κορυφής του Λυσίου Μεγάρου που χάριξε το δρόμο και στη συνέχεια ε, το Δεκέμβριο του 2014 στον πρόεδρο Μάκη Σάρτ και ε, ακολούθησε και επόμενη με συμμετοχή πάνω από 100 προσώπων, αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, ε, κοινωνία των πολιτών. Κάποιο αναφέρθηκε στην κοινωνία των πολιτών. Είναι πάρα πολύ σημαντική για να εκτελούνται όλε οι αποφάσει. Ε, διάφοροι ερευνητέ κλπ. Έγινε επίση μέγα λόγο για τι νέε προκλήσει στην ασφάλεια στην Αφρική, μια ολοκληρωμένη στρατηγική κατά τη τρομοκρατία, αλλά συζητήθηκε επίση και η μεταρρύθμιση ε, του κλάδου της ασφάλειας, καταπολέμηση της πειρατείας στη θάλασσα, του ηλεκτρονικού εγκλήματος ή και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας. Απευθύνθηκε έκκληση για να ενισχυθεί ε, η ε, ομάδα των κρατών G5 Σαχέλ στις 16 Δεκεμβρίου στο Βέλγιο. Θα γίνει μια συζήτηση και παρακαλώ να μας υποστηρίξετε για να καταπολεμήσουμε την τρομοκρατία στην ε, Αφρική ε, θα πρέπει να έχουν καλύτερη εκπαίδευση και κατάρτιση δυνάμεις ασφαλείας. Ε, είναι πολύ σημαντικό ατού το να ξέρει κανείς το έδαφος, το ανάγλυφο για να τους κυνηγήσει σε διάφορα βουνά μέχρι τα τελευταία λιμέρια που κρύβονται. Επίσης, οι πρώοι μαχητές που ιτήθηκαν σε διάφορα θέατρα μάχης βρίσκουν καταφύγιο τώρα σε αφρικανικές χώρες που δεν έχουν υπηρεσίες πληροφοριών ε, αποτελεσματικές. Γι' αυτό χρειάζεται μεγάλη συνεργασία μεταξύ των χωρών που ε, είναι γειτονικέ και μεταξύ των διαφόρων δυνάμεων ασφαλείας. Στην ασφάλεια έχει πολύ μεγάλη σημασία εμείς οι βουλευτές να ασχοληθούμε για να εκπροσωπούνται περισσότερο οι γυναίκες εκεί έτσι θα μειωθεί ε, αδιαμφισβήτητα ε, ο αριθμός των σεξουαλικών επιθέσεων και των βιασμών κατά των γυναικών. Συχνά η απόγνωση ε, στέλνει την νεολαία μας στη μετανάστευση. Νέοι 18 με 40 ετών συχνά μπαίνουν σε κάτι σαπιοκάραβα και πολλές φορές με γυναικόπαιδα μαζί τους. από τότε που περιορίστηκε αυτό, οι διακινητές, οι ασυνείδητοι, ε, στη Λιβύη τους πουλούν ως σκλάβους. Αυτά είναι απαράδεκτα πράγματα ε, στον 21ο αιώνα. Πού είναι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια. Άκουσα χθε την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να λέγει, κατά τα εγγένεια, η βουλευτής, δεν θυμάμαι ποιος το είπε, ότι θα υπάρξει αποστολή της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Λιβύη. Και θα ήθελα να απευθύνω έκκληση, όχι έκκληση, επιθυμία είναι και ε, το δικό μας κοινοβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συμμετέχουμε σε αυτή την αποστολή. Πολύ σημαντικό γιατί είμαστε εκπρόσωποι ε, λαών. Θα πρέπει ακριβώς να κάνουμε τη φωνή μας να ακουστεί για να μην ξαναδούμε τέτοια φαινόμενα. Ο κόσμος εμάς έχει εμπιστευτεί τη μοίρα του και οι Ευρωπαίοι και οι Αφρικανοί. Η ίδια απόγνωση λοιπόν οθεί τους νέους μας στα ακραία φαινόμενα στην ρίζοσπαστικοποίηση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδοτεί πολλά έργα στην Αφρική, το είπε προηγουμένως η κυρία Γκόμες, στην ασφάλεια, άμυνα, ανθρώπινα δικαιώματα, ανάπτυξη της νεολαίας και των γυναικών κλπ. Αλλά αυτό που λείπει είναι η παρακολούθηση και αξιολόγηση. 50 εκατομμύρια απελευθερώθηκαν προφ σφατά για τη χρηματοδότηση των ομάδων G5 Σαχέλ για να λειτουργήσουν. Και ε, χαιρόμαστε γι' αυτό, αλλά ως βουλευτές θα πρέπει να έχουμε ενημέρωση για να βλέπουμε πώς γίνεται ε, ο έλεγχος ε, της κυβέρνησης και αν διαχειρίζεται καλά τα κονδύλια. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα πρέπει να βασιστεί στο Παναφρικανικό Κοινοβούλιο που εκπροσωπεί τους λαούς της Αφρικής που θα συνεργαστεί με τα 55 κράτη-μέλη της Αφρικανικής Ένωσης για να υπάρχει αποτελεσματική παρακολούθηση. Το σημαντικότερο πρόβλημα για τις αφρικανικές χώρες που εμποδίζει την ανάπτυξη είναι η ασφάλεια, γιατί χωρίς την ειρήνη πού να τη βρει την ανάπτυξη. Οι ομάδες, μάλλον οι δυνάμεις του ΟΗΕ ε, έχουν παρουσία σε πολλές χώρες αλλά δεν είναι πάντα αποτελεσματικές. Το Μάλι η Μινούσμα είναι κάτι ε, το οποίο όλο και περισσότερο βρίσκει τον πληθυσμό απέναντι. Μόνο στις πόλεις ε, είναι η μήνουσμα στον ΚΑΟ α πούμε τις προάλλες ο κόσμος σκοτωνόταν και ήταν ε, παρόν ο ΙΕ και δεν έκανε τίποτα και ποιος κάνει το λαθρεμπόριο ναρκωτικών κάποιοι ε, πρώην στρατιωτικοί δήθεν ε, με τα μεληθέντες, το ξέρουν και οι, ομάδες, οι μονάδες Μπαρκάν και οι ΙΕ και οι πάντες, κανείς δεν κάνει τίποτα. Ας ασχοληθούμε λοιπόν εμείς για να εφαρμόζονται σωστά τα ψηφίσματα του ΙΕ για να βγει ο κόσμος από αυτή την κατάσταση και η Αφρική ειδικότερα. Θα πρέπει να αγωνιστούμε κατά της ριζοσπαστικοποίησης. Οι γυναίκες θα πρέπει να συμμετέχουν περισσότερο σύμφωνα με το ψήφισμα 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας για να προλαμβάνουμε να ε, ευαισθητοποιούμε τη νεολαία γιατί αν δεν ε, εμπλακούν οι γυναίκες δεν υπάρχει καμία ε, προοπτική εγώ είμαι πρόεδρος του κόκους του Παραφρικανικού Κοινοβουλίου της ομάδας ε, αυτή που ασχολείται με τις γυναίκες και προσπαθούμε κυρίω να εστιάσουμε στην πρόληψη και της τρομοκρατία αλλά και ε, για τι εκλογές. Γιατί οι εκλογές είναι επίση πηγή ε, σύγκρουσης. Κάθε φορά που βλέπουμε κάτι που κινδυνεύει να πάει στραβά στέλνουμε αποστολέ στον Μπουρούντι ε, στη λαϊκή δημοκρατία του Κονγκό και πάει λέγοντας για να δούμε τι συνέβη. Η πρόληψη όμως είναι το καλύτερο φάρμακο για να εξαλείψουμε αυτή την ε, ανασφάλεια που επικρατεί παγκοσμίω. ευχαριστώ για την ευγενή σας προσοχή. Ο κύριος Ντόνζον, τελευταίος. Ε, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε θέλω να κάνω κάποια εισαγωγικά σχόλια πριν κάνω ερώτηση στα μέλη του πάνελ, γιατί αυτό είναι. Ακούω κάποιες ομιλίες που λένε ότι για όλα αυτά με εμείς. Ε, ας συνετιστούμε λίγο. Τα όπλα, η οικονομία, τα λεφτά, η μετανάστευση, για όλα αυτά με εμείς, οι Ευρωπαίοι. Είτε το ένα κάνουμε είτε το άλλο, πάντα εμείς φταίμε. Όλα τα στραβά ψωμιά. Και αυτό είναι και προσβλητικό για τους Αφρικανούς μας φίλους. Γιατί αν κοιτάμε μόνο ως μετανάστευση το μέλλον της Αφρικής, δεν μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορούν να μείνουν στις χώρες τους και να τις αναπτύξουν. Αυτά τα βρίσκω και περιφρονητικά και σοκαριστικά. Ποια είναι η νόμιμη μετανάστευση. Αυτό είναι χήμερα και μύθος απόλυτος. Απόλυτος. Πώς θα καταπολεμήσουμε τους διακινητές μόνο με νόμιμες οδούς και τις ροές πώς θα τις απορροφήσουμε. Δεν πρόκειται όλες. Υπάρχουν λύσεις κάπως πιο... Υπάρχουν νόμιμοι διάδρομοι. Δεν πρόκειται ως διαμαγές να φύγει. Ή θέλετε να, να, να υποδεχτείτε όλα τα εκατομμύρια των μεταναστών εδώ. Όλα αυτά δεν είναι καθόλου βιώσιμα. Λοιπόν, α πρετανεύσει λίγο η, λογική. Καλό είναι να αγανακτούμε και να διαρριγνύουμε τα ημάτια μα συναισθηματικά. Κυρία Γκόμες, μην μιλάτε, λέει η Πρόεδρο, θα σας δώσω το λόγο μετά. Μην διακόπτετε τον ομιλήτη. Έλεγα λοιπόν, για να συζητήσουμε με τα μέλη του πάνελ. Γιατί προσκαλέσαμε κόσμο για να συζητήσουμε μαζί του. Ε, ήταν καταπληκτικές οι παρουσιάσεις και θα ήθελα να το σχολιάσω και να κάνω ερωτήσεις. Έχω πολύ συγκεκριμένες ερωτήσεις. Πρώτη ερώτηση. Για την αποστολή UCAP στον Ήγυρα. Πριν από λίγα χρόνια την είχαμε επισκεφθεί εκεί. Και μας λέγανε ήδη ε, οι ντόπιοι εκεί στον Ήγηρα ότι έκανε πολύ καλή δουλειά. Αλλά ένα από τα προβλήματα ήταν ότι η κατάρτιση ήταν γενετικά ποιοτική πλην όμως Στη συνέχεια δεν ε, υπήρχε παρακολούθηση από πλευρά εξοπλισμού. Το εγκληματολογικό, η σήμανση, ε, οι υπηρεσίε τη αστυνομία ε, είχαν εκπαιδευτεί, αλλά η εκπαίδευση αυτή τελικά ήταν μια τρύπα στο νερό, γιατί δεν του δίναμε τον εξοπλισμό που χρειάζονται. Ε, σήμερα λοιπόν υπάρχει αυτός ο υλικοτεχνικός εξοπλισμός που θα έρθει να υποστηρίξει την εκπαίδευση που τους έχουμε κάνει. Και λέω για τις ευαίσθητες ψυχές ότι δεν μιλάω για όπλα εδώ, ε, για διακίνηση κλπ. Μιλώ για επιστημονική και εγκληματολογική υπηρεσία της αστυνομίας που χρειάζονται κάποια ε, υλικοτεχνική υποδομή. Πολύ ωραία αυτά που είπατε κύριε Ανακόβο, πάρα πολύ σωστά. Γνωρίζουμε πολύ καλά ότι στην περιφέρεια του Αγκαντές κυρίως η διαχείριση των λαθρεμπορίων και των διακινητών είναι οικονομικό μοντέλο και αυτό δεν ανάγεται στον πόλεμο της Λιβύης. Σας μην γελιόμαστε. Αυτό είναι μια πρόφαση ε, που μας βολεύει για να πούμε ότι τα προβλήματα ήρθαν το 2011. Λυπάμαι, αλλά η αστάθεια στο Μάλι είναι δεκαετιών. Βεβαίως, ενισχύθηκε με τη Λιβύη, αλλά δεν πυροδοτήθηκε από εκεί η κρίση στην Αφρική νότιος της Σαχάρας, απλώς επιδεινώθηκε. Ε, ο σπόρος της αστάθειας υπήρχε από καιρό και σωστά το είπε ο κύριος Λέμποβιτς, ότι οι αφρικανικές χώρες διαχειρίστηκαν με διαφορετικό τρόπο την αστάθεια αυτή. Η συμπερίληψη που έκανε ο Νίγηρας χωρίς αποκλεισμούς ε, μπορεί να μην είναι ε, πλήρη, το είπατε και εσείς ο ίδιος, αλλά λειτουργεί καλύτερα από τα όσα γίνονται στο Μαλί. Επίση θα πρέπει να καταλάβουμε ότι η αδυναμία των ε, αρχών του Μαλί να λύσει τα προβλήματα στο Βορρά ευθύνεται περίπου εξίσου με τον πόλεμο στη Λιβύη. Το οικονομικό μοντέλο λοιπόν βασίζεται σε διάφορα λαθρεμπόρια, όχι μόνο διακίνηση ε, μεταναστών στον Καντές. Υποκατάστατο πώς θα βρούμε οικονομικό και κοινωνιολογικό ε, σχετικά μέσω πρόθεσμα, όχι μέχρι αύριο, αλλά ε, για να τους αποσπάσουμε τους ανθρώπους αυτούς, να τους αποτρέψουμε από αυτό το οικονομικό μοντέλο που είναι ιδιαίτερα διεστραμμένο ε, και ε, κακό. Για το G5 του Σαχέλ όλοι χαιρετίζουμε, χαιρετίζουμε αυτή την προσπάθεια. Βεβαίως χρειάζονται περισσότερα χρήματα οι αρχές της τοπική αυτοδιοίκησης για να καταπολεμήσουν την αστάθεια. Όλα αυτά είναι πολύ καλά και σωστή λύση. Πλην όμως εκφράζεται έντονη αμφιβολία ως προς τη δυνατότητά τους να ανταποκριθούν και την ηλική αλλά και τη δυνατότητα συνεργασίας μεταξύ τους, γιατί ο καθένας έχει άλλη ατζέντα. Πώς το βλέπουν τα μέλη του πάνελ και ποιες θα πρέπει να είναι οι ζώνες προτεραιότητας με τις οποίες πρέπει να ασχοληθεί. Ευχαριστώ. Η Άννα Γκόμες, έχεις το λόγο ε, προσωπικού αλλά πάρα πολύ σύντομο στα γαλλικά. Θέλω κάτι να διευκρινίσω όταν μιλώ για την ελεγχόμενη μετανάστευση. Αυτό εννοώ, ελεγχόμενη μετανάστευση. Να έχουμε νόμιμες οδούς και ασφαλείς έτσι ώστε ο κόσμος που θέλει ε, να ε, ζητήσει και έχει θεμητά ε, αιτήματα και λόγο να έρθει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και ταυτόχρονα μόνο έτσι θα υπάρξει διακυβέρνηση και εκεί, στην Αφρική. Για να παραμείνουν στην Αφρική, εκεί που είναι οι άνθρωποι και εκεί που θέλουν να παραμείνουν, αν υπάρχουν συνθήκες αξιοπρέπειας και ανάπτυξης και να ζουν αξιοπρεπώς. Thank you. Σας ευχαριστώ. Τώρα θα ήθελα οι πανελίστες μας να απαντήσουν στις ερωτήσεις ε, που ετέθησαν και από τους Ευρωπαίους και τους Αφρικανούς βουλευτές. Ξεκινάμε και πάλι με τον κύριο Φερσμέσεν, τον αναπληρωτή διοικητή ε, μίστρετ των επιχειρήσεων. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Ευχαριστώ για τις συγκεκριμένες ερωτήσεις που αφορούσαν εμένα. Ναι, λίγες ήταν αυτές οι οποίες αφορούσαν συγκεκριμένα την αποστολή. χάρηκα που συμμετέχουν εδώ πέρα και οι βουλευτές από τα Αφρικανικά Κοινοβούλια. Βλέπουμε εδώ πέρα ακριβώς την πολυπλοκότητα και το μέγεθος των προκλήσεων, την περιφερειακή διάσταση επίσης, που είναι πολιτικής φύσης και αυτό ισχύει γενικώ και για το ζήτημα της μετανάστευσης και νομίζω ότι η Πατή εκπρόσωπος εξέθεσε το όραμά της Ε, χτες ε, στο Κοινοβούλιο. Να σας ε, πω κάτι. Η αποστολή αυτή στον Ήγυρο, στον είναι μία αποστολή, μία από τις τρεις αποστολές που έχουμε στην περιφέρεια. Εμείς θέλουμε ακριβώς να υλοποιήσουμε την έντολή μας με βάση αυτά τα οποία έχουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε συνεργασία με άλλους με τον ΟΗΕ και τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης. Για να σας δώσω ένα παράδειγμα, η αποστολή συμμετέχει σε αυτό το οποίο ανέφερε ένας ομιλητής στο λεγόμενο Συμβούλιο Ειρήνης ε, για να βρεθούν ακριβώς εναλλακτικές ε, στον κλάδο της ε, λαθροδιακίνησης και ακριβώς ε, προσπαθούμε να διευκολύνουμε την παρουσία μας εκεί επί τόπου. Το ένα θέμα είναι ότι εμείς είμαστε πολιτική αποστολή και με τους ανάλογους φορείς ε, συνεννοούμεθα. Βεβαίως η πραγματικότητα είναι ότι μιλάμε για διοκτικές αρχές και η επιβολή του νόμου γίνεται μόνο από τις ένοπλες δυνάμεις σε κάποιες ε, περιοχές. Συνεργαζόμαστε λοιπόν με τις ένοπλες ε, δυνάμεις ε, για ζητήματα και ανθρωπίνων δικαιωμάτων με στόχο όμως να μπορούν προσεχώς και οι πολιτικοί φορείς, οι μη στρατιωτικοί φορείς να αναλάβουν το έργο της επιβολής ε, του νόμου. Αν έχει βελτιωθεί η κατάσταση, νομίζω ότι έχει βελτιωθεί η κατάσταση και στη διαλειτουργικότητα και στις ικανότητες. Μιλάω για τα περιφερειακά επιχειρησιακά κέντρα, αλλά ναι, παραδέχομαι ότι έχουμε πολύ δρόμο ακόμα μπροστά μας. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Στους πρώτους 8 μήνες του 2017 οι δυνάμεις ασφαλείας συνέλαβαν 1091 μετανάστες που είχαν εγκαταληφθεί στην έρημο από λαθροδιακινητές Τι, πώς αντιμετωπίζουμε λοιπόν το ζήτημα είναι μη εκτελεστική η αποστολή δεν τα κάνουμε εμείς λοιπόν και ενισχύουμε βεβαίως την ικανότητα των τοπικών φορέων. Έχουμε βεβαίως και την διαχείριση. Απλά πράγματα. Τι κάνουμε σε έναν τόπο εγκλήματος, ε, έρευνες, ε, προανακρίσεις. Ε, έχουμε τις κοινέ ομάδες έρευνας που εκπαιδεύσαμε τους Νιγηριανούς συναδέλφους και κατάφεραν να διαλύσουν διάφορα κυκλώματα διακίνησης για το θέμα του εξοπλισμού, κύριε Ντανζάν. Η σχέση των αποστολών ΚΕΠΑ και εξοπλισμού δεν ήταν ποτέ ευθεία, δεν ήμασταν εμείς στο έργο της ανάπτυξης, όμως έχει υπάρξει μια σχετική ανάπτυξη και αυξήθηκε ο προπολογισμό από τα 3,1 εκατομμύρια πέρσι σε 5 εκατομμύρια φέτο για να αντιμετωπίσουμε και το ζήτημα του εξοπλισμού και έχουμε και διμερεί επαφέ ακριβώ για το θέμα του εξοπλισμού και τη εκπαιδευτέλωση για το G5, το G5 είναι στρατιωτική φύσεως, οπότε δεν θα πω τίποτα γι' αυτό, αλλά είμαστε έτοιμοι και στον Νίγηρα και μέσω της αποστολής στο Μαλή να στηρίξουμε το αστυνομικό κομμάτι τους ε, προγραμματιζόμενης αυτής δύναμης ε, G5. Σας ευχαριστώ. Θα ήθελα τώρα να δώσω τον λόγο στον πρόεδρο, τον κύριο Ανάκο, τον Περιφερειάρχη. Ε, ευχαριστώ, πρόεδρε. Ο κύριος Ανάκο. Παρακολούθησα τόσα δεν ήταν απλώς αγορεύσεις. Όσα ακούσαμε σήμερα ε, πρέπει να απαντήσω στις σχετικές ερωτήσεις. Κάποιος? Αναφέρθηκε στο πώς θα σταματήσουμε πιο αποτελεσματικά τους ε, διακινητές και αναφέρθηκε κάτι σαν ε, οικονομική ενίσχυση, αποζημίες, πολύ επικίνδυνη αυτή η ιδέα. Είπαμε ότι έχουμε εκπαίδευση στρατού και ε, αστυνομικών, τα είπε ο εκπρόσωπος της UCAP. Θα πρέπει να μην φέρουμε σε απόγνωση τον πληθυσμό. Να σεβαστούμε τον κόσμο. Αυτό είναι η πρώτη μας δουλειά. Τώρα για τους διακινητές. Ποια πρόσωπα είναι αυτά. Ποιοι κάνουν αυτή τη δουλειά. Στο Άγκαντες, στην περιφέρειά μου, είναι κάποια πρόσωπα που ποτέ δεν θεωρούνται εγκληματίες. Τα έχουμε συζητήσει αυτά με την ε, κυβέρνηση. Τα συζητήσαμε με την αντιπροσωπεία της Ένωσης. Όχι. Δεν είναι εγκληματίες. Είναι νέοι. Που κέρδαν τους ομίλους από τον τουρισμό που δεν υπάρχει πια. Και από τον 10 ο αιώνα έχει ξεκινήσει η μετανάστευση. Οπότε αυτοί οι άνθρωποι βρίσκονται στο σταυροδρόμι. Και πάντοτε οργανώναν τα καραβάνια, τη, τη, τη, τη διάσκηση της ερήμου, τη μεταφορά. Τα είπαμε στην κυβέρνηση του Νίγηρα και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και όλοι οι αιρετοί άρχοντες του Αγκαντές μαζευτήκαμε και διατυπώσαμε πρόταση προς την κυβέρνηση της χώρας και προς την Ένωση. Θα πρέπει να δώσουμε εναλλακτικέ σε αυτούς τους νέους. Για να σταματήσουν αυτή τη δουλειά. Να είναι σε αυτά τα δίκτυα της λαθροδιακίνησης. Γενικά, οι νέοι αυτοί άνθρωποι είναι παλαιοί πολεμιστές όταν είχαμε την επανάσταση στο παρελθόν. Άρα Και είπαμε σε αυτούς τους νέους. Ε, από σήμερα και πέρα είναι παρανομή η μετανάστευση, άρα προσέχτε. Γιατί αν η αστυνομία σας πιάσει τα πράσα, θα σας συλλάβει όπως προβλέπει ο νόμος. Ε, είπαμε αντεπιχειρήματα για τον νόμο, κάναμε κάποιους ε, απολογισμό των επιπτώσεων και τελικά η εναλλακτική είναι το να ασχοληθούν με άλλη δραστηριότητα αυτοί οι άνθρωποι. Υπάρχει ένα πρόγραμμα να δούμε τι θέλουν να κάνουν για να σταματήσουν αυτή τη δραστηριότητα. Κάναμε προτάσεις. 7.000 ήρθαν σε επαφή μαζί μας. Πολλοί από αυτούς έχουν μαγαζιά, εστιατόρια. Πρόκειται για ένα ολόκληρο κύκλωμα. Δεν είναι ότι ασχολούνται αυτοί μόνο με την διακίνηση. Καλά υπάρχουν και εγκληματίες. Αλλά δεν θα πρέπει τους βάζουμε όλους στο ίδιο καλάθι. Πρόκειται για μια ολόκληρη οικονομία στην περιφέρεια. Θα πρέπει να αντικατασταθεί αυτή η δραστηριότητα με μια άλλη. Άρα να τους κάνουμε πρόταση, να τους δώσουμε ένα πρόγραμμα αλλαγής και σε όλους τους εταίρους είπαμε τις ε, ιδέες μας. Έχουν 6 μήνες, 7 μήνες. Περιμένει ο κόσμος, περιμένει αυτοί οι νέοι. Οπότε θα ξαναγυρίσουν στη δραστηριότητα εκείνη. Θα πρέπει επομένως να αποφύγουμε, να αποτρέψουμε αυτό να έχουν μπροστά τους ε, αυτή την, την επιλογή. γιατί τώρα θα αρχίσει η πραγματική διακίνηση. Και μια που είναι τόσο ευάλωτα τα πράγματα, τους ελκύουν και οι τρομοκράτες. Ε, δίπλα στη Λιβύη είμαστε και καταλαβαίνετε ότι μπορεί να στρατολογηθούν αυτοί οι άνθρωποι. Είμαστε δίπλα στο Μαλί. Έτσι δυστυχώς είναι τα πράγματα και γι' αυτό και κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου ούτως ώστε ταχύως να βρεθεί μια λύση. Και εμείς και οι εταιροί μας κάνουμε ό,τι μπορούμε. Είναι κατεπήγον το θέμα. Κάτι θα πρέπει να γίνει επιγόντως. Τώρα, για να πάμε στο θέμα της Λιβύης. Δεν είναι η Λιβύη το πρόβλημα των προβλημάτων. Πάντου υπάρχουν συγκρούσεις, προστριβές, πόλεμοι στην Αφρική. Εκεί αποτύχαμε. Δηλαδή, δεν λάβαμε υπόψη της κοινότητας, τους λαούς, της τον κόσμο. Άρα, θα πρέπει οι κυβερνώντες στο μέλλον να είναι πιο δίκαιοι με το λαό τους, με τη χώρα τους. Γιατί εκεί που υπάρχει η επανάπτυξη βρίσκουν έδαφος οι τρομοκράτες. Να, τι γίνεται στη Βόρεια Νιγηρία. Εκεί. Αυτές οι απομακρυσμένες περιοχές. Α, ρωτήστε τους βουλευτές του Παναφρικανικού Κοινοβουλίου είναι οι πανάπτυκτες απομακρυσμένες γεωγραφικές περιοχές αυτές. Όχι, δεν φταίει το Ισλάμ όπως είπε κάποιος. Το θέμα είναι οικονομικό, είναι η απελπισία των μειονοτήτων σε κάποια κράτη. Οπότε βρίσκει έφορο έδαφος η τρομοκρατία. Στο Νίγηρα το αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα με υπεύθυνο τρόπο και σε εμά στο βορρά. Είναι η πιο ευάλωτη περιοχή ο βορράς, εκεί που είχαμε συγκρούσεις και με την αποκέντρωση ανέλαβε τις ευθύνες του κόσμου για να διαχειριστεί τα του οίκου του. Άρα για όλα τα προβλήματα θα πρέπει κανείς να αναρωτηθεί. Γιατί, γιατί δεν υπάρχει τρομοκρατία στο Αγκάντες, αλλά Μπορεί να στατολογηθεί ο κόσμος για τρομοκρατία. Όμως το αποφύγαμε αυτό. Έχουμε θωρακίσει τον κόσμο. Τους δώσαμε τις ευθύνες τους κατά κάποιο τρόπο. Και έτσι δεν έχουμε τρομοκρατία. Άπαξ και εφόσον εμπιστεύονται την αποκέντρωση, άπαξ και εφόσον οι εταίροι μας μας υποστηρίζουν Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε κύριε Λέη Πρόεδρος και να δώσουμε τώρα τον λόγο στον ε, κύριο Λέμποβιτς από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων. So Σας ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί ο χρόνος πιέζει. Σύντομα. Ε, θα μέση θέση για, τους, ε, για τις νόμιμες διόδους μεταναστευσής είναι πολιτικά ε, ευαίσθητο. Εντάξει, δεν νομίζω ότι είναι κατακριτήριο να λέμε ότι ο κόσμος θέλει να μεταναστεύσει για κάποιους λόγους και πάλι πέραν από το οικονομικό ε, και ιστορικά συνέβαινε. Αυτό το οποίο λέγαμε και αυτό το οποίο έχω πει εγώ και στα γραπτά μου είναι ότι πρέπει να υπάρξει ένας συνδυασμός κάποιας νόμιμης μετανάστευσης στην Ευρώπη και ενθάρρυνση της περιφερειακής μετανάστευσης. Έτσι θα έχουμε ε, και κάποιες νομικές διατάξεις αλλά και οικονομικά προγράμματα που θα πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση όχι μόνο αναπτυξιακά αλλά προγράμματα για βιομηχανία για σε διάφορους κλάδους, στην Αλγερία, στο Μαρόκο, ως μέρος της πολιτικής στρατηγικής μας, για να ενθαρρυνθεί η περιφερειακή μετανάστευση. Είναι πολιτική η πρόκληση, αλλά ταυτόχρονα είναι μία δυνατότητα για να αντιμετωπίσουμε αυτά τα ζητήματα. Το πρόβλημα τώρα είναι ότι με την τρέχουσα πίεση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σταματήσει και η περιφερειακή μετανάστευση εντός της ΕΚΟΒΑΣ που είναι η περισσότερη μετανάστευση ε, πλέον καθίσταται πιο δύσκολη. Και αυτό είναι το αποτέλεσμα της πίεσης της Ένωσης και πρέπει να το θυμόμαστε. Ότι ε, αυτά τα οποία κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει αντίκτυπο σε αυτές τις περιοχές, ειδικά στον ε, πληρώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση 40% νομίζω του προϋπολογισμού της χώρας. Οπότε δεν είναι ότι δεν έχει καμία επιρροή. Αλλά αυτό σημαίνει ότι όταν ασκεί η πίεση η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κυβέρνηση δεν έχει άλλη επιλογή από το να ανταποκριθεί. Και αυτό έχει συνέπειε βέβαια σε ολόκληρη τη χώρα και ιδιαίτερα στο βορρά. Και αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκόμε είναι σημαντικό. Πρέπει να υπάρξουν πιο συνεκτικά προγράμματα επανένταξης στο παρελθόν τα προγράμματα αφορούσαν την ηγεσία των εξεγέρσεων στη δεκαετία του 90 και πιο παλιά αλλά δεν έκανε τίποτα για τους μαχητές ε, από εκεί και κάτω και μετά ποιοι ήταν οι κλάδοι που μπορούσαν να κατευθυνθούν. Τουρισμός, ε, εμπόριο ναρκωτικών, ε, λαθροδιακίνηση. Όταν υπάρχει δουλειά κάτι κάνουν. Τώρα που δεν υπάρχει τουρισμός και καταστέλλεται η λαθροδιακίνηση υπάρχουν λίγες επιλογές. Ο τουρισμός είναι πρόκληση γιατί προφανώς ε, κανένας κανένα κράτος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν θέλει να απαχθούν οι υπηκόοι του στον Βόρειο Νίγηρα. Ε, βεβαίως υπάρχει και ένα θέμα εδώ γιατί το πρόβλημα είναι ότι τα κράτη-μέλη δυσκολεύουν και τους πολίτες τους να ταξιδέψουν εκεί και λένε όλη η χώρα, όλο το Σαχέλ είναι κόκκινη ζώνη και δεν μπορεί ο κόσμος να λάβει και τις σχετικές αποφάσεις ε, και υπάρχει τουρισμός αυτή τη στιγμή στον Βόρειο Νίγηρα. Δεν είναι διαφημίζεται αλλά υπάρχει. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι ε, έχουν κάνει τουρ ε, με πλήρη ασφάλεια. χρειάζονται κατάλληλε διασυνδέσει και οι κατάλληλη υποστασία, αλλά υπάρχουν κάποιε δυνατότητε. Και για το θέμα των ε, G5 εγώ ήμουν μία από τις εναλλακτικέ φωνές, θα έλεγα, για τις δυνατότητες. Νομίζω ότι μπορεί να ωφελήσει οριακά με την έννοια ότι δεν είναι κακή η περιφερειακή ολοκλήρωση, η διαλειτουργικότητα στα σύνορα δεν είναι κακή, αλλά γενικά μία από τις ανησυχίες μου είναι ότι όπως όλοι εκεί πέρα προσπάθησαν να κάνουν τους G5 προτεραιότητα στην περιοχή. Βλέπουμε και κάποιες προτεραιότητες στην εντολή των G5 που δεν είναι πολύ ρεαλιστικές. Μιλάμε π.χ. για την ένταξη εκεί πέρα και της μετανάστευσης, ασφάλειας αυτών των ζητημάτων. Δεν θα τα αντιμετωπίσει, δεν μπορεί να τα αντιμετωπίσει. Έχει και το οργανωμένο έγκλημα ως εντολή. Είναι παράλογο, για να μιλή κανείς για το σχόλιο που έγινε για την αστυνομία και τις δυνάμεις ασφαλείας του Νίγηρα που διέλυσαν τέτοια δίκτυα διακινητών. Θα ήθελα περισσότερες πληροφορίες γιατί κατά την εμπειρία μου και με τις συζητήσεις που είχα εγώ στον Νίγηρα τα δίκτυα τα οποία διαταράσσονται είναι στοχευμένα δίκτυα. Κάποια διαταράσσονται και κάποια άλλα λειτουργούν ανεμπόδιστα είναι κομμάτι ακριβώς της διαδικασίας που ανέφερα στις παρατηρήσεις μου, αλλά α, εντάξει, υπάρχει κάποια πρόοδος, αλλά να ξέρουμε και το τι γίνεται όταν μιλάμε για διάλυση δικτύων. Μπορούμε να πούμε ότι το εμπόριο ναρκωτικών δεν έχει μειωθεί στο Σαχέλ ε, και κανείς ε, και η αστυνομία δεν μου έχει πει ότι το εμπόριο έχει αλλάξει σε κάποιες περιπτώσει έχει αυξηθεί και είναι και αυτό ένα σοβαρό ζήτημα ε, δεν πρέπει να μας παραπλανούν σχόλια που λένε ότι διαλύονται τα δίκτυα κτλ να μιλάμε και για την οικονομία, ε, ναι, είναι σημαντική, αλλά για εμένα από αυτά πολλά από αυτά τα ζητήματα είναι και πολιτικά και πρέπει να τα δούμε σφαιρικά. Και η τελευταία μου έκκληση είναι ότι άκουσα κάποιε παρατηρήσει σήμερα ότι φαίνεται ότι ακόμα και σε βασικά ζητήματα υπάρχει ανάγκη πληροφόρησης και ανάλυσης. Εντάξει, βεβαίως εγώ τι θα έλεγα, αυτό θα έλεγα, αλλά ως ερευνητής Νομίζω ότι πρέπει να υπάρχουν και οι συζητήσεις υψηλού επίπεδου που έχουμε εδώ, αλλά και συζητήσεις ει βάθο ε, που ελπίζω θα βοηθήσουν την χάραξη πολιτικής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δυστυχώς δεν έχουμε χρόνο για άλλη συζήτηση. Πρέπει να περάσουμε στο επόμενο θέμα της ημερησίας διάταξης. αξιονόματος ολόκληρης της υποεπιτροπής θα ήθελα να ευχαριστήσω τους πανελίστες μας ε, και ειδικά τους Αφρικανούς εταίρους μας ε, που εμπλούτησαν την συζήτηση αυτή. Σας ευχαριστώ και σας καλώ να αναφωνήσουμε να χειροκροτήσουμε τους ε, συναδέλφους μας. Ευχαριστώ.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 Oh, thank you very much Κυρίες και κύριοι, καθίστε παρακαλώ, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε τη συζήτηση για το επόμενο θέμα. Με ιδιαίτερη χαρά και τιμή πέρασαμε στο επόμενο θέμα και θα σας συστήσω τα ξέχοντα μέλη του πάνελ με στρατιωτική αποστολή ε, και ΠΑ για την στήριξη της μεταρρύθμισης του τομέα ασφαλείας στο Ιράκ. Και πάλι καλωσορίζουμε τον κύριο Μπέρτ Βερσμέσεν, αναπληρωτή διοικητή μη στρατιωτικών επιχειρήσεων και προσωπάρχη της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης, καθώς επίσης και τον κύριο Καουά Χασάν, ήδη γνωστό μας, γιατί είχαμε την ευκαιρία να συνομιλήσουμε μαζί του και να ακούσουμε την παρουσίασή του και στο παρελθόν. Ο κύριος Χασάν είναι διευθυντής στο πρόγραμμα Μέσα Ανατολής και Βόρειας Αφρικής το East West Institute. Λοιπόν, θα ακούσουμε πρώτα τον κύριο Χασάν να μας κάνει μια επισκόπηση γενική της ε, παρούσης κατάστασης ασφαλείας ε, στην χώρα και τις πολιτικές εξελίξεις. Θα μας ε, γράψει με βάση την ευρύτερη κατάσταση ασφαλείας στην περιοχή και μετά θα επικεντρωθούμε στις ε, επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Αποστολής εκεί. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you very much, um, Good morning. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σας. Αξιότιμα μέλη της Επιτροπής, κυρίες και κύριοι. Ε, σας ευχαριστώ και πάλι για την καλοσύνη που είχατε να μας προσκαλέσετε πάντα με μεγάλη μας τιμή ερχόμαστε για να μοιραστούμε τις σκέψεις του East West Institute μαζί σας και προσβλέπω σε μια πολύ γόνιμη συζήτηση μαζί σας. Την περασμένη φορά που απευθύνθηκα ήταν πριν από ένα χρόνο γιατί ανέτρεξα στην ατζέντα μου. Νομίζω 28 Νοεμβρίου ήτανε. Και τότε λοιπόν σας ανέλησα την ε, κατάσταση ε, ε, ασφαλείας στη μάχη της Μοσούλης κατά του ISIS. Σήμερα μου ζητήσατε να σας αναλύσω γενικότερα τις εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις του Ιράκ και τη μακροπρόθεσμη ανασφάλεια και ένταση μετά την επέμβαση των ΗΠΑ, το ISIS, το κουρδικό, την επέμβαση ε, του περιφερειακών δυνάμεων, ε, βασικές μεταρρυθμίσεις που χρειάζονται για τη σταθεροποίηση της χώρας κλπ. Όλα αυτά θα προσπαθήσω ε, όσο γίνεται να τα καλύψω μέσα σε ένα τέταρτο. Πολλά είναι τα θετικά που συνέβησαν ως αλλαγές από την περασμένη φορά που συναντηθήκαμε. Αλλά παραμένουν τα βασικά προβλήματα και βασικές προκλήσεις. Τι έχει ακριβώς αλλάξει τότε Πρώτον, οι Ιρακινές δυνάμεις ασφαλείας και ένοπλες δυνάμεις, η αντιτρομοκρατική, η Πεσμεργά, η αστυνομία, όλοι αυτοί με την υποστήριξη της Διεθνούς Συμμαχίας επέτυχαν μια μεγάλη νίκη κατά του ISIS. Η τρομοκρατική οργάνωση εκθιώθηκε από τις περισσότερες βασικότερες πόλεις που κατήχε το 2014 και ε, μετέπειτα. Αυτή είναι μια μαζική στρατιωτική νίκη που αξίζει την υποστήριξη και την αναγνώριση της διεθνούς κοινότητας. Αλλά και το κόστος είναι αμέτρητο. Πριν σας δώσω μερικά στοιχεία, αριθμητικά θα ήθελα να τονίσω ένα σημείο. Παρά αυτή τη στρατιωτική νίκη, είναι πολύ σημαντικό και πάλι να τονίσουμε ότι ο πόλεμος κατά του ISIS δεν έχει ακόμα τελειώσει. Ούτε πρόκειται να τελειώσει προσεχώς. Ακόμα και αν καταλάβουν και την ύπεθρο οι Ιρακινές δυνάμεις τις επόμενες εβδομάδες και μήνες. Είναι ασυνείδητη ε, τρομοκρατική οργάνωση, εφάνταστη, πολυμήχανη, ε, ευκίνητη, ευέλικτη, που κάθε φορά επανεφευρίσκει τον εαυτό της για λόγους που θα σας αναλύσω στη συνέχεια είναι τεράστια η κοινωνική, ανθρώπινη και ηλική καταστροφή. Είναι δύσκολο να σας δώσουμε αριθμητικά στοιχεία για τις απώλειες και τους νεκρούς από το 2014, αλλά σύμφωνα με τα επίσημα κοινά στοιχεία, οι νεκροί και οι τραυματίες άμαχοι είναι 15 με 20.000 στην περιοχή γύρω από τη Μοσούλη. Οι μισοί ε, ε σκοτώθηκαν στη Μοσούλη και μάλιστα χιλιάδες ε, εκτιμώνται οι αγνοούμενοι. Από τις 15 Νοεμβρίου περίπου 3 εκατομμύρια είναι οι εσωτερικά εκτοπισμένοι. Και συνολικά με τους πρόσφυγες 1,9 εκατομμύρια και 183.000 οι Κούρδοι που έφυγαν από το ε, Κυρκούκ και το Τούθ Χουρμάτου μετά την ανάκτηση των πόλων αυτών. Από τις 15 Νοεμβρίου, σύμφωνα με το Διεθνή Οργανισμό, 2,6 εκατομμύρια 150 δισεκατομμύρια δολάρια θα κόστιζε η ανασυγκρότηση. Αναεπαρχία το κόστος αυτό κυμαίνεται, αλλά το συνολικό είναι δυσθεώρητο. Πάνω από 120 δισεκατομμύρια ε, θα είναι ε, και το χρέος του Ιράκ. Παρά την ε, παραγωγή που, που έχει 130 δις θα είναι μέχρι τα τέλη του έτους, παρά τη συνεχιζόμενη σταθερή παραγωγή πετρελαίου. 4,5 δισεκατομμύρια βαρέλια παράγουν την ημέρα, αυτό αναμένεται να αυξηθεί κατά 10% και να γίνει 5 δις εκατομμύρια ε, βαρέλια. Είναι τεράστια λοιπόν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει και η μεγαλύτερη ερώτηση είναι μπορεί η Ιρακινή κυβέρνηση και τα βασικά πολιτικά κόμματα να μεταφράσουν την ε, στρατιωτική νίκη σε μια βιώσιμη πολιτική επιτυχία ή μήπως μετά από λίγο χρόνο θα ξαναπέσει το Ιράκ ολόκληρο στον ε, φαύλο κύκλο της βίας στην οποία μπατα βία. Βεβαίως οι Ιρακινοί ηγέτες θα πρέπει να απαντήσουν σε αυτή την ερώτηση και να λύσουν τα βασικότερα προβλήματα. Πλην όμως η διεθνή κοινότητα και η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί και οφείλει να διαδραματίσει επικοδομητικό σημαντικό ρόλο στην υποστήριξη της ανοικοδόμησης ε, και της πολιτικής και της ουσιαστικής φυσικής για να γίνει το Ιράκ από θέατρο πολέμων ε, διατυπροσώπων σε μια δομή χωρίς αποκλεισμούς και να είναι με τον εαυτό του συμφιλειωμένο με τους γείτονες ε, και τον κόσμο όλο. Μπορεί να επαναλαμβάνομαι, αλλά αυτό είναι αναπόφευκτο και κρίσιμο να το λέμε. Το ISIS είναι η απόρρια και όχι η αίτια, η αιτία συγγνώμη, των δεινών που υφίσταται το Ιράκ. Και δεν υπάρχει περίοδος μετά το ISIS τώρα. Θα πρέπει λοιπόν να καταλάβουμε και πολιτικά και ουσιαστικά και να μιλούμε ότι μετά το 2003 ε, απέτυχε το κράτος. Τα σημερινά προβλήματα στη Μέση Ανατολή και τη Βόρεια Αφροκή έχουν να κάνουν με την πολιτική τάξη μετά το 2003, όχι μετά το 2014, όπου προέλασε ο ISIS. Χωρίς να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, το πολιτικό σύστημα ε, που ε, ανελήφθηκε από το 2003 μετά την πτώση του Σαντάμ, απέτυχε να κάνει ένα κράτος χωρίς αποκλεισμούς που να βασίζεται στην ηθαγένεια, στην ίση κατανομή και επιμερισμό ε, του πλούτου και της εξουσίας με λογοδοσία. Αυτό ισχύει και για τη Βαγδάτη και για το Ερμπίλ. Ενδεχομένως ένας από τους πιο ε, ορατούς δείκτες για την αποτυχία των κυβερνήσεων και στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ είναι ότι μετά από 14 χρόνια είναι τεράστια τα προβλήματα που έχουν οι Ιρακινοί πολίτες για τις βασικές καθημερινές υπηρεσίες. Υπάρχει διαφθορά παντού στην κορυφή και μάλιστα το Ιράκ δεν είναι και φτωχή χώρα. Με δύο λόγια, το πολιτικό σύστημα είναι μπλοκαρισμένο. Οι πολιτικοί ηγέτες που κυβερνάνε από το 2003 αναπαράγονται και η εμπιστοσύνη των πολιτών στα πολιτικά κόμματα και στους θεσμούς του κράτους μειώνεται δραματικά και ε, ε, στις κουρδικές περιφέρειες και στο Ιράκ. Αντί να δίνουν το παράδειγμα και να έχουν μια ηγετική ε, στάση και να επηρεάζουν παντού οι μεγάλοι πολιτικοί ηγέτες, αναλώνονται σε ρητορικές, διχαστικές, εκταριστικές, περιχαρακώνονται στο θρησκευτικό τους ε, και το κοινωνικό περιβάλλον και ε, μιλούν για εξωτερικές παρεμβάσεις. Πώς θα σπάσει αυτό λοιπόν, για να αλλάξουν τα πράγματα, να αντιστραφεί η τάση. Βεβαίως η Ιρακινή κοινωνία δεν είναι παθητική. Έχει δείξει άνευ ανθεκτικότητα κατά ε, της δικτατορίας του Σαντάμ Χουσέιν αλλά και κατά του αυταρχισμού και της διαφθοράς των ελίτ μετά του Σαντάμ και κατά της βαρβαρότητας του Άισις. Πολιτικός κατακαιρματισμός ε, είναι καθημερινό φαινόμενο παντού και στο Κουρδιστάν και στο υπόλοιπο ε, Ιράκ. Ο κατακαιρματισμός βεβαίως δεν είναι κατά ανάγκη αρνητικός. Μπορεί να σημαίνει δημοκρατία αλλά μπορεί να οδηγήσει και σε ταραχές και σε εμφύλιο πόλεμο. Αυτό λοιπόν που χρειαζόμαστε ποιο είναι. Επειδή η δυναμική επιτόπου ε, είναι ρευστή ε, και πολιτικά και κοινωνικά, θα πρέπει να καταλάβουμε ότι υπάρχει μεγάλη δυναμική ε, και εξελίσσεται το τοπικό περιβάλλον. Πιο μακροπρόθεσμα η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να αντιμετωπίσει τα αίτια της κρίσης κυρίως τη διαφθορά στην κορυφή του κράτους, ε, πολιτικές λειτουργίες, οικονομικά προβλήματα και δημοκρατικό έλλειμμα ε, του κράτους μετά το 2003. Ε, η στρατηγική της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσε να ασχολείται με την ανθρωπιστική βοήθεια μένα, αλλά αυτό δεν αντικαθιστά το πολιτικό κενό. Χρειάζεται ένα πολιτικό πλαίσιο γενικό και μια στρατηγική που θα κάνει στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ μεταρρυθμίσεις ουσιαστικέ, όχι καλοπιστικές. Επίσης, η διαρθρωτική βοήθεια θα πρέπει να έχει στόχο να διαλύσει τις πολιτοφυλακές και κάποιες άτακτες ομάδες που υποτίθεται ότι είναι ε, στα χέρια διαφόρων υπουργείων στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ, αλλά ουσιαστικά ε, είναι ε, κάποια σχήματα ελεγχόμενα προσωπικά από κάποιους ηγέτες. Θα πρέπει να ενισχυθούν οι ένοπλες δυνάμεις και ε, το Ιράκ και η Πεσμεργά των Κούρδων. Η καταπολέμηση της διαφθοράς είναι τεράστιο ε, έργο, αλλά επειδή ο κόσμος ε, έχει απογοητευτεί, η κοινωνία των πολιτών πιέζει για διαφάνεια και λογοδοσία. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υπολογίζει στην υποστήριξη των Ιρακινών. Ωστόσο αυτό χρειάζεται μια στρατηγική μακροχρόνια προσέγγιση έτσι ώστε το σύστημα να μην αναπαράγεται. Η καταπολέμηση της διαφθοράς από την κορυφή προς τη βάση χρειάζεται ισχυρή αντιμετώπιση θεσμούς μη κομματικούς, ανεξάρτητους, ε, ικανούς, κεντρική τράπεζα και λοιποί θεσμοί θα πρέπει ε, να μην έχουν πολιτικές παρεμβάσεις ούτε κομματικές παρεμβάσεις. Ε, θα πρέπει να τα πούμε ξεκάθαρα αυτά ε, και στην κυβέρνηση και στα πολιτικά κόμματα του Ιράκ. Επίσης, εκστρατείες, συνειδητοποιήσεις για το τι κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, η κυβέρνηση του Κουρδιστάν έχασε 50% των, ε, ε, της επικράτειας που ήταν αφιλεγόμενη και το Κυρκούκ και 60% των εισοδημάτων μετά το ψήφισμα. Πάνω από 183.000 κυρίως Κούρδοι έχουν εκτοπιστεί εσωτερικά και έχουν πάει σε περιφέρειες που ελέγχονται από τους Κούρδους. δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να σταθεροποιήσουμε και να ενισχύσουμε μια μη δημοκρατική κυβέρνηση στο Κουρδιστάν. Και η κουρδική κοινωνία έχει απογοητευτεί με την ελίτ και την αντιπολίτευση και δεν υπάρχει και καμία προοπτική για να λυθεί το σημερινό τους πρόβλημα οικονομικό και πολιτικό. Άρα θα έχουμε ένα Κουρδιστάν μετά το ISIS και ένα Ιράκ μετά το ISIS που θα χαρακτηρίζεται από την ε, άνοδο ε, ακραίων ιδεών θρησκευτικών και μη και περαιτέρω παρέμβαση τοπικών ε, δυνάμεων, περιφερειακών παραγόντων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να βοηθήσει ε, και στα πολιτικά κόμματα να προχωρήσουν σε ελεύθερες και δίκαιες εκλογές. Αυτό ισχύει και για την κυβέρνηση. Μήπως να τα πείτε λίγο πιο αργά για να σας προλαβαίνουμε γιατί έχουμε κάποια προβλήματα ταχύτητας με τη διερμηνή. Λοιπόν, πιο ε, σημαντικό είναι ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να υποστηρίξει νέα κόμματα, κοινωνικά κινήματα, δημοκρατικά και πολιτικά ε, στη Βαγδάτη και στο Ερμπίλ που ανθίστανται στην κυβέρνηση και έχουν αναγνωριστεί από τον τοπικό πληθυσμό. Με δίκαιες, ελεύθερες, αξιόπιστες εκλογές του χρόνου, εάν προχωρήσει αυτό, ο σημαντικό βήμα στην καταπολέμηση ε, αυτών των νέων πολιτικών και κοινωνικών κινημάτων για να υπάρχει ένα σύστημα θεσμικό και όχι καταφυγή στη βία και δεχομένως επαναστατικές κινήσεις και πράξεις. Τελευταίο, τα εσωτερικά διαθροτικά προβλήματα του Ιράκ δεν μπορούν να ειδωθούν ε, σπασμένα από την ε, γειτονία, την ευρύτερη. Ένα ασθενές Ιρακινό κράτος καλεί ε, εξωτερικές επεμβάσεις που ε, αποσταθεροποιεί ολόκληρη την περιοχή και πρόσφατα είδαμε προσέγγιση με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα και τη Σαουδική Αραβία. Αυτή είναι μια εξέλιξη ευπρόσδεκτη που θα πρέπει να εθαρρυνθεί. Μετά την ήττα του ISIS, η Ιρακινή κυβέρνηση θέλει να παίξει ένα ρόλο καταπραϊντικό ε, στην ε, μείωση των εντάσεων μεταξύ του Ιράν και της Σαουδικής Αραβίας. Το Ιράκ λοιπόν θα πρέπει να κάνει τη μετάβαση τώρα από ένα θέατρο ε, πολέμων δια σε μια δομή που θα υποστηρίζει ιδέες που θα έχουν στόχο να δημιουργηθεί η εμπιστοσύνη η οικονομική αλληλεξάρτηση μεταξύ των χωρών συνεργασίας του κόλπου με κοινά σχέδια ανοικοδόμησης των περιοχών που έχουν απελευθερωθεί από το ISIS και γενικότερα να υπάρξει ένα πλαίσιο για τη συνεργασία. Το Ιράν, η Τουρκία και άλλες χώρες της περιοχής μπορούν και οφείλουν να συμμετέχουν στην οικονομική συνεργασία εκεί. Μόνο μια, ένα Ιράκ ε, δίκαιο, σταθερό και ένα σύστημα ασφαλείας γενικότερο στην περιοχή μπορεί να εγγυηθεί ένα Ιρακινό κράτο χωρίς αποκλεισμού με σταθερότητα. Ένα τελευταίο θέλω να πω για το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωση στη βελτίωση ε, των σχέσεων ε, μεταξύ ε, της Βαγδάτης και, και των κουρδικών κομμάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συνομιλεί και με το Ερμπίλ και με τη Βαγδάτη και θα πρέπει να χρησιμοποιήσει αυτή τη δυνατότητα που έχει για να προωθήσει ενδεχομένως ε, και να φιλοξενεί συνομιλίες του KRG και της Βαγδάτης ιδιαίτερα μετά από όσα συνέβησαν στις 16 Οκτωβρίου και τις επόμενες ημέρες. Είναι ιστορική, πιστεύω, αυτή η εταιρεία για να διευθετηθούν όλα τα εκκρεμούντα θέματα ε, και ως προς τις εξουσίες και προς τις επικράτειες που είναι αφισβητούμενες. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Indeed, Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Τώρα να δώσουμε λόγο στον κύριο Μπέρτ Φερσμέσεν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι βουλευτές, η συζήτηση οπωσδήποτε είναι επίκαιρη και για την αποστολή καθώς χθες το βράδυ στην Βαγδάτη είχαμε τα εγγένεια με τους Ιρακινούς ε, συνομιλητές μας και όπως είπα χθες ο διοικητής των πολιτικών επιχειρήσεων είναι εκεί με την επικεφαλή της αποστολή. Θα έλεγα κάτι για το ευρύτερο πλαίσιο, αλλά νομίζω ότι ακούστηκαν ήδη όσα πρέπει να ακουστούν. Εγώ θα πω δύο πράγματα μόνο. Πρώτον, ότι τον Ιούνιο φέτος ε, το Συμβούλιο Εξωτερικών ζήτησε από την Κομισιόν και την Υπατεκπρόσφα να αναπτύξει μια στρατηγική για το Ιράκ, η οποία καταρτίζεται και δεύτερον, όταν δείτε την χώρα, βλέπετε ότι εγκρίθηκε μια στρατηγική Εθνικής Ασφαλείας. Από το Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας ε, τον Οκτώβριο του 2016 έχουμε ένα πρόγραμμα μεταρρύθμισης του κλάδου της ασφαλείας ε, από το ίδιο Συμβουλίο τον Ιούλιο φέτος ε, και με βάση αυτό το πλαίσιο και της στρατηγικής και του σχεδίου εφαρμογής οι αρχές του Ιράκ ζήτησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση να βοηθήσει στην μεταρρύθμιση των δυνάμεων ασφαλείας. Ε, το τονίζουμε γιατί δεν έχουμε παντού ε, ένα σχέδιο και μια στρατηγική εφαρμογής αλλά και την βούληση της κυβέρνησης να συνεργαστεί μαζί μας. Και βεβαίως ε, το Ιράκ τώρα και η διεθνής ε, κοινότητα πρέπει να αντιμετωπίσουν τους νέους ε, κινδύνους ε, μετά από την ήττα βέβαια του Ισλαμικού κράτους που έχει βεβαίω κάποιες αποχρώσεις. Είπαμε ότι ήμασταν έτοιμοι κατόπιν ετήματος των Ιρακινών αρχών να αναπτύξουμε μια ομάδα συμβούλων και βοήθειας. Είχαμε αναπτύξει την, ε, το σχετικό σχέδιο τον Ιούλιο και εγκρίναμε και το επιχειρησιακό σχέδιο και τη νομική βάση, την απόφαση δηλαδή, για να συσταθεί αυτή η δύναμη και 17 Νοεμβρίου η βασική ομάδα και κάποια στελέχη κλειδιά αναπτύχθηκαν στην Βαγδάτη και βεβαίως οι υπόλοιποι θα ξεκινήσουν την επόμενη εβδομάδα από τις Βρυξέλλες. Έχουμε λοιπόν την πτυχή της ασφαλείας και τις πολιτικές πτυχές. Έχουμε λοιπόν στρατηγικές συμβουλές ε, για την εφαρμογή των πολιτικών πτυχών την στρατηγική SSR, την οποία ανέφερα, και στρατηγικές αντιτρομοκρατίας και οργανωμένου εγκλήματος. Δεύτερον, συντονισμός και συνεργασία που περιλαμβάνει και συντονισμό και διαχείριση της κοινή γραμματείας και τέλος στρατηγικός σχεδιασμός και ανάλυση κενών για να βρούμε ευκαιρίες για πιθανή μελλοντική στήριξη στην εφαρμογή των στρατηγικών αυτών. Και βεβαίως εστιάζουμε στην εφαρμογή του σχεδίου μεταρρυθμίσεων Ε, την αντοχή των θεσμών, αντιτρομοκρατία, πρόληψη τρομοκρατίας και καταπολέμηση βίαιου ε, εξονισμού και τέλος ε, διαστάσεις του οργανωμένου εγκλήματος περιλαμβανομένου του εγκλήματος που αφορά την λαθροδιακίνηση αρχαιοτήτων. Επίσης βεβαίως προσπαθούμε να δούμε το τι θα γίνει σε σχέση με το μέλλον, να βρούμε ευκαιρίες για μελλοντικές έμπλοκες ε, ε, της Ένωσης είτε μέσω του ΚΕΠΑ είτε με κάποιον άλλο τρόπο. Τώρα ε, αυτή τη στιγμή έχουμε έδρα στην Βαγδάτη, στην κόκκινη ζώνη, στο ξενοδοχείο Βαβυλώνα. Αποτελείται από 50 άτομα με έναν προπολογισμό 14 εκατομμύρια ευρώ. Επικεφαλής είναι ένας υψηλόβαθμος γερμανός αστυνομικός Μάρκους Ρίτερ λέγεται με το και βεβαίω ένα σημαντικό στοιχείο θα είναι η συνεργασία με άλλους ε, οργανισμούς, συγκεκριμένα τον ΟΗΕ και το πρόγραμμα ανάπτυξης του ΟΗΕ. και πρέπει ακριβώς να υπάρξει συνοχή μετά όσα κάνει ο Ιε. Προφανώς αυτό είναι στην στρατιωτική πλευρά και έχουμε και άλλους ε, εταίρους ε, ε, και υπάρχει και η Παγκόσμια Συμμαχία κατά του Ισλαμικού κράτους. Αυτά λοιπόν ως έτσι, μια βασική δράση εστιάζουμε στη μεταρρύθμιση των σωμάτων ασφαλείας ε, και περιοριζόμαστε στην Βαγδάτη, θα είναι δύσκολο να έχουμε αποτελέσματα τόσο γρήγορα. Για την ώρα η εντολή είναι για ένα έτος. Και βεβαίως ε, έχουμε ακριβώ ε, την είμαστε περήφανοι για το ότι καταφέραμε να αναπτυχθούμε μέσα σε ένα μήνα ε, να αναπτύξουμε την βασική ομάδα και ελπίζουμε να είμαστε επιχειρησιακοί πριν το τέλος του έτους για να ξεκινήσουμε να έχουμε αποτελέσματα. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε κύριε, κύριε Φερμέσεν και ευχαριστούμε για όλα αυτά που είναι χρήσιμο που μας εξήγησε. Ο κύριος Ντόνσον πρέπει να φύγει, οπότε να δώσουμε σε εσά το πρώτο το λόγο. Ευχαριστώ πρόεδρε. Συνάδελφοι, δυστυχώ πρέπει σε λίγο να φύγω. Ε, Βεβαίω και πρόσεξα ότι είπε ο κύριο Χασάν για τι ανάγκε που υπάρχουν, τι ρόλο μπορεί να παίξει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Συμφωνώ βέβαια με την ανάλυση του και προσ... να προσέξουμε να μην έχουμε ψευδεστήσει όσον αφορά το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για κάτι τόσο περιπλοκό, δηλαδή όπως το θέμα της ε, σταθεροποίησης του Ιράκ, γιατί όπως μας υπενθυμίσατε το βασικό πρόβλημα από το οποίο εκπηγάζουν όλα τα άλλα όσον αφορά την διακυβέρνηση, την σωστή διακυβέρνηση, είναι, είναι θέμα πολιτικής, είναι θέμα της καρδιάς τη Ιρακινής κοινωνίας και των διαφόρων επιμέρους κοινοτήτων και η Ευρωπαϊκή Ένωση φοβάμαι δεν μπορεί να πειράσει και πολύ όλες αυτές τις σημαντικές μεταβλητές. Ίσως μπορεί σε έναν μικρό βαθμό και να μην ξεχνούμε ότι υπάρχουν όλες αυτές οι τεκτονικές πλάκες στην ε, περιοχή σε σχέση με την Τουρκία, σε σχέση με τις ΙΠΑ. Ε, ε, πολύ σχετική η δύναμη επιρροής μας. Οπότε συμφωνώ με το θεματολόγιο, αλλά φοβάμαι ότι από μόνοι μας, αλλά ακόμα και χέρι-χέρι με άλλους, δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά. Ε, βλέπουμε πόσο δυσκολία έχουμε. Δεν μπορούμε να επηρεάσουμε ούτε καν τις χώρες της ε, γειτονίας μας που είναι υποψήφιες για προσχώρηση. Ε, τότε τι, τι, τι να, τι θεωρούμε ότι να κάνουμε σε σχέση με το Ιράκ. Δεν λέω να είμαστε απόντες. Αυτό θα ήταν ακόμα χειρότερο. Κάπου μεταξύ του όλα και του τίποτα. Άρα, πού το πάω. Στο εξής. Ως ερώτηση, ως παρατήρηση. Ακριβώς για την ασφάλεια και την αποστολή σας. Ε, βέβαια, και η ασφάλεια στο Ιράκ είναι ένα συνοθήλευμα από νόμιμες δυνάμεις, από πολιτοφυλακές, από τα αφεντικά, κάποιους ισχυρούς ε, και από τη μία μεριά ε, έχουμε δίπλα όλους αυτούς τους πολλούς ε, Αμερικανούς συμβούλους και από την άλλη τους επίσης πολλούς Ιερανούς συμβούλους. Οπότε το πρόβλημα είναι τι θα γίνει στο Ιράκ. Τι θα κάνουμε, θα κάνουμε αυτό που κάναμε στην, στο Αφγανιστάν χωρίς και πολλή επιτυχία επί τη βάση των στρατηγικών συμβουλών όλα αυτά που ξεκίνησαν θεωρητικά πολύ καλά σε υψηλό επίπεδο αλλά επί επιτόπου τα πράγματα ήταν πολύ χλωμά και ως προς τους Αφγανούς και ως προς το τι έγινε με τον ΝΑΤΟ. Άρα μην κάνουμε τα ίδια και στο Ιράκ. Ε, να μην τα κάνουμε επειδή πρέπει να τα κάνουμε. Για να λέμε ότι τα κάναμε γιατί να λέμε ότι είμαστε παρόντες. Βεβαίως και πρέπει να υπάρχει εκεί η παρουσία μας και δεν ξέρω αν ε, αυτού του είδους η αποστολή είναι το πιο δόκιμο μέσο. Έχω πολλές αμφιβολίες γιατί τα έχω ξαναδεί και αλλού. Είπαμε για Νίγηρα, είπαμε για Μαλή και εκεί υπάρχουν επιπτώσεις, εκεί επηρεάζουμε γιατί έχουμε και τα θέματα της οικονομικής βοήθειας οπότε εκεί έχουμε ρόλο κλειδί. Στο Ιράκ όμως δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο, πρέπει να αποδειχθεί. Θα σε ευχαριστώ κυρία Γκόμες. Σύμφωνο με τις απόψεις του Αρνό Ντονζόν. Πρέπει όμως να σας πω Υπάρχουν πολλές ε, εξηγήσει γιατί δεν έχουμε τόσο στιβαρή παρουσία στο Ιράκ. Είναι γιατί κάποια κράτη-μέλη εκείνα δηλαδή που θεωρούν ότι μπορούν να έχουν και έχουν επίδραση και επιρροή στο Ιράκ, δεν θέλουν Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτό εξηγεί γιατί. Στις επιχειρήσεις κατά του Ισλαμικού κράτους, πολλές φορές είπα στην κυρία Μογκερίνη γιατί η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν στέκεται πρωτοπόρα και ηγέτιδα, μα γιατί δεν το θέλουν τα κράτη-μέλη. ήθελαν να είναι παρόντα τα μέλη. θέλανε το συντονισμό. Ναι, ναι, θα πρέπει και να υπάρχει η παρουσία μας. Βέβαια, αυτό είναι μια αρχή. Ε, όχι. Και να απουσιάζουμε. Το 8. Μας στη Και τότε είχαμε την αποστολή της Ένωσης στην Βαγδάτη. Και αυτό έγινε μέσω των Βρετανών, της Βρετανικής Αποστολής. Δεν θα πρέπει να υπάρχουν εγκαταστάσεις για αυτόνομη αποστολή της Ένωσης. Ε, το, το πήγαμε να το κάνουμε, αλλά υπήρχαν θέματα διαχείρισης. Υπήρχε αντίσταση από κράτη-μέλη. Δεν είχαμε αυτονομία. Το 2007-2008 πήγα εκεί και ο εκπρόσωπος της Ένωσης εκμεταλλεύτηκε το δικό μου ταξίδι για να πάει γιατί ποτέ δεν είχε βγει από την Βαγδάτη και με την ευκαιρία της δικής μου επίσκεψης πήγε στη Συρία για πρώτη φορά πήγε στους Κούρδους είναι θέμα αυτονομίας, αυτοτέλειας, πολύ σημαντικό Τώρα με το Brexit ακόμα χειρότερα. Άρα η αποστολή στη Βαγδάτη να έχει αυτονομία, αυτό τέλειο. Και να μπορεί να πάει παντού στη χώρα, χωρίς πρόβλημα και κυρίως στις κουρδικές περιοχές, ακριβώς για να αναλάβει αυτό το ρόλο που μας εξηγήσατε και συμφωνώ. Μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να το κάνει αυτό. Ιδίω μια που είναι τόσο περίπλοκες οι σχέσεις Βαγδάτη-Ερμπίλ. Φοβάμαι αυτό που φοβάται και ο Αρνό. Μην καταλήξουμε να κάνουμε τα ίδια, να μην κάνουμε τίποτα όπως το Αφγανιστάν. Θα πρέπει να είμαστε εδώ πιο φιλόδοξοι. Κάπως να χειριστούμε. Ε, τα πράγματα και όχι μόνο την ασφάλεια σαν αστυνομική, πολύ πιο φιλόδοξη να είμαστε και είναι και το θέμα του εκδημοκρατισμού, όπως είπατε. Και στη Βαγδάτη και στις κουρδικές περιοχές. Γιατί ακριβώ αυτό ήταν το πρόβλημα τα τελευταία χρόνια. Ήταν μπλοκαρισμένο το κοινοβούλιο, ε, δεν μπορούσε ο κόσμος να μιλήσει ελεύθερα. Εδώ μπορούμε να παίξουμε ένα σημαντικό ρόλο. Ναι, να συνεργαστούμε με τον ΟΗΕ, αλλά να κάνουμε και εμείς κάτι. Να μην είμαστε υποχείρια. Μην έχουμε κάποιες δομές που στερούνται στρατηγικής. Τελευταία φορά που πήγα, πέρσι στη Βαγδάτη. Όχι, όχι, πήγα στο Ερμπίλ πήγα. Για να δω τι γίνεται με την ανθρωπιστική βοήθεια. Και είδαμε ότι δεν υπήρχε σύνδεσμος, δεν υπήρχε συνεννόηση. Και ακόμα και στο πλαίσιο της Ένωσης μεταξύ υπηρεσιών ανάπτυξης και ανθρωπιστικής βοήθειας. να θέμα μόνο κατά επίγουσα τη ανθρωπική βοήθεια, θέμα του να βοηθήσουμε για την παιδεία, τα σχολεία κλπ. Να, τι γίνεται και στου κόλπου τη Ένωση. Άρα πρέπει να έχουμε στατικό σχεδιασμό και θα πρέπει πραγματικά να ασχοληθεί η κυρία Μογκερίνη, να χρησιμοποιήσει τα εργαλεία που έχουμε και το Κοινοβούλιο. Νομίζω ότι μπορεί να παίξει κάποιο ρόλο και θυμάμαι ότι από τότε που ξεκίνησε η αντιπροσωπή για το Ιράκ έκανα και την έκθεση του 8 και μέχρι τώρα η αντιπροσωπεία δεν έχει μπορέσει να ταξιδέψει, να πάει στη χώρα. Γιατί δεν, δεν έχει δοθεί το πράσινο φως ο πρόεδρος ασφάλειας εδώ από το Κοινοβούλιο. Ε, αυτό είναι, είναι αδιανόητο. Είναι δική μας αρμοδιότητα. Η αντιπροσωπεία μας που τόσους και τόσο οι καλέσει από το κοινοβούλιο του Ιράκ, Ιρακινούς, Κούρδους λοιπά να μην μπορεί να πάει εκεί. Αυτό θα πρέπει να αλλάξει. Πρόεδρε, μιλήστε με τον πρόεδρο, τα Δεν είναι δυνατόν να συνεχιστεί αυτή η πολιτική και εμείς θα πρέπει κάτι να κάνουμε σε σχέση με την αποστολή. Και σε συνεννόηση με τους ε, κοινοβουλευτικούς Ιρακινούς συναδέλφους και Κούρδους. Ε, ευχαριστούμε. Καλά, θα το λάβουμε αυτό υπόψη, λέει η πρόεδρος. Και τώρα ο κύριος και έχει το λόγο. Δύο τι να, να σας αναφέρω. Πρώτον, η θέση των χριστιανών στο Ιράκ. Πώς το βλέπετε, τι γνώμη έχετε για το θέμα ασφαλείας αυτών Ποιες θα ήταν οι καλύτερες πολιτικές συνθήκες από πλευράς του πώς περνάνε αυτοί οι άνθρωποι, αυτές οι κοινότητες, γιατί ξέρουμε ότι τα τελευταία 15 ετία έχουν υποστεί πολλά. Άρα, για πετε μου σε σχέση με την πολιτική κατάσταση, μπορείτε να μας τα πείτε εις βάθος, γιατί μας μιλήσατε για ανθρώπινα δικαιώματα, μας μιλήσατε για την δυναμική δημοκρατία, αλλά θεωρούσαμε ότι ε, αυτά ήταν το φάρμακο για κάθε πρόβλημα της χώρας. Όμως με δεδομένο αυτόν τον φατριασμό, ε, την πολλαπλή διάσπαση της κοινωνίας, τι θα ήταν το καλύτερο πλευρός πολιτικών εξέλιξεων για τις μειονότητες και πιο συγκεκριμένα για την χριστιανική μειονότητα επίσης. Δεύτερον, Ίσως ε, είναι πολύ πρόημα αυτό που λέω, αλλά αν μπορείτε, πέστε μας για τις επιπτώσεις αυτής της τραγωδίας. Δηλαδή της ύπαρξης της δράσης του Ισλαμικού κράτους. Πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα Ξέρουμε ότι και στη Συρία υπάρχουν τέτοιοι τρομοκράτες και αλλού. Οι συνέπειες αφορούν όλη την περιοχή. Πώς το βλέπετε. Ίσως με την πτώση του Ισλαμικού κράτους, ίσως καταπέσουν και οι παραφιάδες του. Γιατί έτσι λειτουργεί το σύστημα Περμούη. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Κοιτάξτε, ήθελα να κάνω κάποιες ερωτήσεις. Συμφωνώ με τον κύριο Χασάν ε, ότι πρόκειται για ένα αποτυχημένο κράτος που δεν ξεκίνησε το 2013. Ήταν καταστροφική η διαχείριση της ε, εισβολής. Κατά την άποψή μου αυτή ήταν ε, παράνομη και αυτά που ακολούθησαν. Αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι Κάποια στιγμή θα φτιάξουν στρατό εκεί, ακόμα και αν είναι ομοσπονδιακό το κράτος. Ένοπλες δυνάμεις εθνικές θα υπάρχουν και μετά από την ε, απόλυτη αποτυχία της μονομερούς κήρυξης ανεξαρτησίας ε, του Κουρδιστάν. Ε, δεν υπήρξαν αιματηρές ε, μάχες για την ανάκτηση των εδαφών, αλλά η κατάσταση είναι δύσκολο να λυθεί. Το ίδιο ισχύει και με την περιφέρεια Αλάμπαρ, που είναι Σουνίτες ιδιαίτερα μετά την καταστολή του 2011 με 2013, που οδήγησε στο γεγονός να πέσουν στην αγκαλιά του Άισις πολλοί Σουνίτες εθνικιστές. Τώρα, Αλμαλίκη, η κοινή κυβέρνηση έχει αλλάξει την ε, αντιμετώπιση του Αλμαλίκη που βασιζόταν στις φατρίες και στις θρησκευτικέ ομάδες. Ε, το Ιράν ε, συμμετέχει στο Ιράκ. Οι Σιήτες ε, ε, βοήθησαν στην απελευθέρωση της Μοσούλης και υπάρχει και η Χεσμολάχ στο Ιράκ. Ε, ευχαριστώ. Εδώ τελειώνει η λίστα των ομιλήτων. Θα ήθελα να κάνω κι εγώ μια ερώτηση, μου επιτρέπετε, και στους δύο ομιλητές μας. Σε κάποιο βαθμό έχει σχέση και με αυτά που ρώτησε ο κύριος Γιούρεκ. Ίσως από μια διαφορετική σκοπιά στη μεταρρύθμιση ε, του κλάδου σωμάτων ασφαλείας και το πρόγραμμα γίνεται ειδική αναφορά και μέρημνα για το πώς θα επιστρέψουν οι εσωτερικά εκτοπισμένοι και πώς θα τους βοηθήσουν. Εμείς κατανοούμε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα. Ακούσαμε τους αριθμούς. Είναι πραγματικά συγκλονιστική. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχουν οι πολιτικές συνθήκες, ε, αλλά είναι εφικτό κάτι τέτοιο από πλευράς έτσι, δύναμης. Έχει τη δυνατότητα το κράτος να προστατεύσει αυτή την επάνωδο στις Με την αντίστροφη σειρά παρακαλώ πρώτα ο κύριος Βέρσμεσεν και μετά ο κύριος Χασάν. Ευχαριστώ πολύ. Κυρία Πρόεδρε. Ε, λίγα συγκεκριμένα έγιναν. Εγώ θα είμαι ε, ε, περιορισμένη στην απάντησή μου. Λοιπόν, έχουμε 51 υπαλλήλους εκεί, 35-36 είναι οι ε, διεθνείς υπάλληλοι και οι υπόλοιποι είναι ντόπιοι. Είναι προσεκτική, συνετή, σταδιακή η προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα και πώς θα βοηθήσουν. πραγματικά καταλαβαίνουμε τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά... Αυτό αντανακλά και τα διδάγματα ε, που ε, εξήχθησαν από την αποστολή στο Αφγανιστάν. Εγώ διστάζω πάντα να ε, συγκρίνω περιοχές, αλλά στο Αφγανιστάν θυμάστε ότι είχαμε στείλει 200 πρώτα και μετά 400 και είχαμε και μεγάλες φιλοδοξίες και μετά δυσκολευτήκαμε να έχουμε αποτελέσματα επί τόπου όταν γεννήσαμε τόσο μεγάλες προσδοκίες δεν θα συμφωνούσα με τα σχόλια για τη βιωσιμότητα και τα όσα έχουμε επιτύχει, γιατί ως προς την εκπαίδευση η αποστολή είχε αρκετά αποτελέσματα. Επίσης, είναι γεγονός ότι όταν τελείωσε η αποστολή πέρσι, είχε μειωθεί η δυνατότητα ανάπτυξης ε, αστυνομίας για ε, τη φύλαξη της χώρας, γιατί ε, σκοτώνονταν πάρα πολλοί αστυνομικοί κάθε χρόνο και τους χρησιμοποιούσαν ουσιαστικά και ως πεζικό. Τώρα σας είπα ότι στο ξενοδοχείο Μπάμπιλον, στην κόκκινη ε, ζώνη, στεγάζεται η αποστολή μαζί με τη Βρετανική Πρεσβεία, αλλά υπάρχουν σχέδια ή αντιπροσωπεία ε, με την αποστολή. Ε, έχουμε και την ευθύνη να προστατεύουμε το προσωπικό μας και εκτός της πράσινης ζώνης και της κόκκινης ζώνης είναι επικίνδυνο μέρος το Ιράκ και η Βαγδάτη. Για να είμαστε εμείς λοιπόν σε θέση να αναπτυχθούμε χρειάζεται ε, κάποιες προδιαγραφές ασφαλείας. Θα εξακολουθούν αυτές να κυριαρχούν λοιπόν και στο μέλλον και ως προς την επιλογή των ε, τόπων. Ε, για τη συνεργασία με τα Ηνωμένα Έθνη, ε, είμαστε αποτελεσματικοί παντού. Το θέμα δεν είναι να υπάρχει ενιαία διοίκηση, όπως συχνά ακούμε, αλλά ενιαίες προσπάθειες, συντονισμός με άλλους κτλ. Any success that, uh, that we can have. Finally, as to your question, Madam President, σε σχέση με τα όσα ρωτήσατε εσείς κυρία Πρόεδρε για την επιστροφή των εσωτερικά εκτοπισμένων, συγγνώμη, ε, δεν είναι δικό μας πρόγραμμα, είναι ε, ε, άλλοι που έχουν επιφορτιστεί με αυτό. Κύριος Χασάν, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις. Ήταν και κρίσιμες πολλές και επικριτικές. Ε, απαντώ στις ερωτήσεις του κυρίου Ντανζάν, ο οποίος ε, έφυγε δεν συμφωνώ με το πρώτο του σχόλιο ότι η κακή διοίκηση και η έλλειψη δημοκρατίας είναι γενή στην Ιρακίνη κοινωνία. Γιατί αυτό χαρακτηρίζει ε, μια κοινωνία και θεωρητικοποιεί ε, κάποιες πολύ περίπλοκες δυναμικές που αναπτύσσονται. Έχει να κάνει, πιστεύω, με το πολιτικό πλαίσιο και το περιβάλλον και την αποτυχία της πολιτικής τάξης στο διάστημα μετά το 2003 να παράξει όχι μια τέλεια δημοκρατία, αλλά πάνω κάτω μια λογική δημοκρατία. πρέπει τα ανθρώπινα δικαιώματα στοιχειοδός, στην αξιοπρέπεια του κόσμου και να πιστεύει σε μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας. Αυτό δεν έχει να κάνει με την Ιρακινή κοινωνία, αλλά με την πολιτική κουλτούρα εκεί στην περιοχή. Γι' αυτό θα πρέπει να το έχουμε υπόψη, έχει σημασία. Αλλιώς θα χάσουμε ε, την περιπλοκότητα και δεν θα μπορούμε να την εκτιμήσουμε. Δεύτερο, οι εξωτερικοί παράγοντες πάντα ε, καλό είναι να δείχνουν συγκράτηση και ταπεινότητα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είμαστε φιλόδοξοι. Υπάρχει διαφορά που θα πρέπει να γίνεται και συμφωνώ με την κυρία Γκόμες ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει πραγματικά ε, και έχει δυνατότητες να πιέσει. Δεν είμαστε Ηνωμένε Πολιτείε, δεν είμαστε κάποιοι άλλοι, αλλά έχουμε την ήπια δύναμη, έχουμε και εμεί τον τρόπο μα. Έχουμε φήμη, έχουμε εικόνα, κύρο. Γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε ε, όλα αυτά. Είναι μάλλον θέμα πολιτική βούληση. Να είμαστε μετριοπαθεί, αλλά και φιλόδοξοι. Και να χρησιμοποιούμε την ήπια δύναμή μα για να έχουμε θετικές ε, αλλαγές. Τώρα, τώρα είναι η ώρα ε, να δράσει η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δραστηριοποιηθεί εκεί. Να φτάσει στην ε, κοινή κοινωνία και να βρει θυλάκους αλλαγής, όπου να μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει στρατηγικό αποτέλεσμα. Την αλλαγή θα την κάνουν οι ίδιοι οι Εξωτερικοί παραγόντες μπορούν να την υποστηρίξουν, να τη βοηθήσουν, αλλά το σημαντικό είναι μόνοι του το κάνουν αυτό. Ε, επανέρχομαι στο θέμα της Ιρακινής κοινωνίας. Βεβαίως, η πολιτική της ταυτότητας παραμένει σημαντική και θα παίξει ρόλο, αλλά βλέπουμε και μετάβαση από την ταυτότητα σε πολιτική με βάση τα θέματα, από το Κουρδιστάν μέχρι τη Βαγδάτη και άλλες επαρχίες. Ε, η έκκληση για χρηστή διακυβέρνηση είναι μια έκκληση που απευθύνεται από όλες τις κοινότητες και τις συνιστώσεις του Ιράκ για καλύτερες κοινωνικές υπηρεσίες. Όλα αυτά τα θέλουν οι άνθρωποι ολόκληρη της χώρας. Βεβαίως τους μεταχειρίστηκαν οι πολιτικοί ε, ηγέτες και θα το κάνουν και στο μέλλον τις διάφορες κοινότητες ε, φατρίες. Αλλά υπάρχουν και άλλοι που πιστεύουν σε πολιτική με βάση όχι το ποιος είσαι, αλλά τα θέματα. Και εκεί μπορούν να παίξουν αυτή θετικό, θετικό ρόλο. Συμφωνώ με τα σχόλια της κυρίας Γκόμε για την έλλειψη δημοκρατίας ε, στη Βαγδάτη και στις κουρδικές περιοχές. Το συζητήσαμε και προηγουμένως. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο τώρα. Όμως και να διευκολύνει μια ειρηνική μεταβίβαση εξουσίας εντός και εκτός των κομματών μετά, κατά τη διάρκεια των εκλογών και το θέμα των διαφιλονικούμενων περιοχών είναι πάρα πολύ κρίσιμο. Ευρω... Τα Ηνωμένα Έθνη δραστηριοποιούνται εκεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενώσει τις δυνάμεις της απευθύνοντας έκκληση στις πλευρές και κάποιες προσπάθειες διαμεσολάβησης. Δεν λέω να αντιγράφει αυτά που κάνει ο ΙΕ, να, τον υποστηρίζει. Τώρα έχει έρθει η ώρα να ε, αρχίσει μια μεγάλη διπλωματική προσπάθεια για να ε, πάνε σε διαπραγματεύσεις και οι Κούρδοι και οι Βαγδάτοι. Οι Κούρδοι το θέλουν, οι Βαγδάτοι λιγότερο, αλλά αυτό θα αλλάξει. Και εγώ είμαι αισιόδοξο για τα όσα μπορούν να γίνουν. Σε σχέση με τα όσα ρώτησε ο κύριος Γιούρεκ, Υπάρχουν χριστιανοί και άλλες μειονότητες που βρίσκονται σε πάρα πολύ δεινή κατάσταση και ε, η δική μου ανάλυση τι λέγει. Ότι οι χριστιανοί, οι και άλλες μειονότητες θα πρέπει να έχουν την ελευθερία να αποφασίσουν ε, τι παρουσία θέλουν να έχουν. Και στην ε, τοπική αυτοδιοίκηση αλλά και στι συνεννοήσεις για την ασφάλεια. Αλλά αυτό θα πρέπει να είναι υπό την αιγίδα ε, εθνικών αρχών ή περιφερειακών στην περίπτωση των Κούρδων που να έχουν την ικανότητα, τον επαγγελματισμό, να μην έχουμε φατρίες, εθνικές ε, προτιμήσεις τι ένοπλε δυνάμει, αλλά αυτά θα χρειαστούν μια γενιά για να γίνουν. Υπάρχουν στα Σπάργανα κάποιες προσπάθειες. Θα πρέπει να αναδιαρθωθεί ο Ιρακινός στρατός με διαφοροποίηση στην κοινωνία, με επαγγελματισμό. Θέλει χρόνο όμως αυτό και πολύ μεγάλη προσπάθεια, κόπο, συνέχεια και θα χρειαστεί μια γενιά μάλλον. Ε, το θέμα του ISIS και το, το μέλλον του. Το μέλλον του ISIS θα εξαρτηθεί από το μέλλον των πολιτικών της Ιρακινής κυβέρνησης και των περιφερειακών κρατών και των Κούρδων. Όλα αυτά είναι αλληλένδετα θα εξαρτηθεί από το τι θα κάνουν αυτοί οι παράγοντες, αλλά και από τον ίδιο τον Άισις. Χάνει δάφη, η ιδεολογία του όμως ζει και βασιλεύει και θα παραμείνει για καιρό εκεί. Πού θα πάνε? Στην έρημο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Μερικοί στην Ευρώπη και άλλες χώρες και στους εσωτερικά εκτοπισμένους καταβλισμούς. Τρεις είναι οι προορισμοί. Πολύ ανησυχητικό για την έρημο. Έχει αρχίσει σήμερα ο κοινό στρατό επιχείρηση για να καθαρίσει τις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Είναι πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή. Γιατί ε, υπάρχουν υποδομές στην ε, επαρχία του Αμπάρ που είναι πολύ μεγάλη, είναι μεγαλύτερη Ιρανική, Ιρακινή συγγνώμη, επαρχία ε, και στη Συρία. Είναι πολύ δύσκολο να τους βρουν εκεί και χρειάζεται βοήθεια από διεθνείς παράγοντες. Αν είναι δύσκολο το έδαφος Στι γύρω χώρε θα είναι πιο εύκολη καταπολέμηση. Αυτό που με ανησυχεί περισσότερο είναι εσωτερικά εκτοπισμένοι ε, στο Σαλαχεντή, ε, στο Αμπάρ, ε, στη Μοσούλη και έχουν πάει και μέλη του Άισι εκεί στου καταβλισμού. Αυτή είναι η μεγαλύτερη μου ανησυχία. Εκεί χρειάζεται πολύ γρήγορα να υπάρξει μια λογική πολιτική για να μετριαστεί και να περιοριστεί η παρεμφάνιση του ISIS, ε, η αναβίωσή του στους καταβλισμούς των εσωτερικών εκτοπισμένων. Αυτά νομίζω κυρία Πρόεδρε. Έχω απαντήσει τα περισσότερα. Uh, colleagues, uh, I think it was... Συνάδελφοι, νομίζω συζητήσαμε αρκετά, είχαμε μια αρκετά μακροσκελή συνεδρίαση με πολύ ενδιαφέροντα σημεία και στις δύο συζητήσεις θα ήθελα να ευχαριστήσω τα μέλη του πάνελ, ε, τους βουλευτές ε, που έλαβαν το λόγο και συνεισέφεραν σε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση και όπως πάντα ευχαριστώ τη Γραμματεία και τους διερμηνείς. Επόμενη συνεδρίασή μας στις 7 Δεκεμβρίου. Αν δεν υπάρχουν διάφορα, λέτε η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.